Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνεδρίαση. Δεν έχω και μικρόφωνο, δεν ξέρω αν πρέπει να πάω αριστερά, δεξιά. Uh, I am start... Ξεκινάει η συνεδρίαση, αν μπορούμε. I, would like to start the meeting. Good morning, everybody. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και να σας ενημερώσω ότι ως συνήθως η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και το πρώτο θέμα της ημερήσια διάταξης είναι η έγκρισή τη. Δεν είχε ζητήσει κάποιος αλλαγέ. εάν λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα, ε, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης, ε, ανακοινώσεις. Να σας ανακοινώσω πολύ σύντομα κάποια πράγματα για τις συνεδριάσεις και τις συναντήσεις που είχα ε, μεταξύ των δύο συνεδριάσεών μας για το Brexit. Εν τω μεταξύ έγινε αρκετά συνεδριάσεις της ε, διευθύνουσα ομάδα για το Brexit με τον Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίο μα είπε κάποια πράγματα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και σε σχέση με τα όσα σας είπα προηγουμένως δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά αν βασιστώ στα προηγούμενα ε, που μας είχε πει ο Μισελ Μπαρανιέ οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται σε καθημερινή βάση. Ίσως η διαφορά είναι ότι πλέον έχουν ε, γίνει πολύ πιο έντονες οι συζητήσεις για τα θέματα που αφορούν κυρίως ε, τη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας στο νησί, το θέμα των συνόρων δηλαδή και τα δικαιώματα των πολιτών. Και νομίζω ότι το ουσιαστικό το οποίο εκκρεμεί αυτή τη στιγμή και ακόμα δεν έχουμε επαρκή πρόοδο είναι το θέμα της οικονομικής εκαθάρισης. Ε, υπάρχουν κάποιες προσδοκίες τώρα ότι το Δεκέμβριο ο διαπραγματευτής θα μπορέσει να ανακοινώσει ότι έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τίποτα και επίσης ε, αυτό αποτελεί και προϋπόθεση για να δώσει και την ευχή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και να προσφέρουμε και νέες ε, διαπραγματευτικές οδηγίες στους διαπραγματευτές. Ε, εν τω μεταξύ, η Διευθύνουσα Ομάδα του Κοινοβουλίου για το Brexit ε, προετοιμάζει τα επόμενα βήματα. Ξεκινήσαμε κάποιες εργασίες για την πρόταση ψηφίσματος, το οποίο θα ψηφίσει ε, το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Ε, θα γίνει η αξιολόγηση λοιπόν η δική μας για το κατά πόσον έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος και ε, θα προτείνουμε και κάποια θέματα που αφορούν κάποιες αρχές και θέματα οριζόντιας φύσεως που αφορούν το στάδιο 2 των διαπραγματεύσεων και αυτά μπορεί να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, δεν έχει αποφασιστεί. Όσον αφορά τις άλλες συναντήσεις που είχα στο μεταξύ, ε, ε, συνάντησα τον Υπουργό Εξωτερικών για τη Σκοτία, τον David Μάντελ, συζητήσαμε διάφορα θέματα ε, που αφορούν και το Brexit αλλά και τις ανησυχίες μας ε, ως Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων που αφορούν ε, τις αποκεντρωμένες χώρες και κυρίως τη Σκοτία. Αυτά είναι για τη Σκοτία. Θες να μιλήσεις, Τζορτζ, για αυτά. Να πω κάτι τελευταίο στις ανακοινώσεις μου. Αμέσως μόλις ήρθε από το αεροδρόμιο είχαμε μια συνάντηση της Κόζακ η οποία ε, συνάντηση ήταν αρκετά σημαντική και ζωντανή θα έλεγα. Έγινε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και οι ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της Εστονίας, ο Μισελ Μπαρνιέ και οι υποφαινόμενοι ως πρόεδρος της ΑΦΚΟ και ως συνήθως στη συνέχεια Δόθηκε χρόνος ομιλίας ενός λεπτού για τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Συζητήθηκαν κάποια θέματα όπως η ψηφιακή ένωση και η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών. Όλα αυτά πολύ σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν και το Κοινοβούλιο. Ως συνήθως υπάρχει η πρόκληση τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις συνεδριάσεις και θα ήθελα να γνωρίζετε κι εσείς ότι θα πρέπει πάντα να υπάρχει παρουσία των πολιτικών σας ομάδων στη συνεδριάση της ΚΟΖΑΚ. Δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ορισμένες φορές πολύ δύσκολα μπορούμε να πείσουμε συναδέλφου να συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, Αυτό θα μπορούσαμε να το θέσουμε και ως ερώτηση στον κύριο Τίμερμανς, γι' αυτό και το αναφέρω. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισε να συστήσει μια task force για τα θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας και το τελευταίο τμήμα του τίτλου ε, είναι «Doing more with less». Να είμαστε δηλαδή πιο αποτελεσματικοί με λιγότερα και αυτή η task force ε, θα αποτελείται από εκπροσώπους ε, τριών θεσμικών οργάνων. Θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Φρανς ε, Τίμερμανς και αυτή η task force θα αποτελείται από εννέα άτομα και κάλεσε τρεις εκπροσώπους επιτροπής Επιτροπή των Περιφερειών, τρεις εκπροσώπους της ΚΟΖΑΚ, δηλαδή Εθνικά Κοινοβούλια, και όχι εμά ε, σε αυτό το πλαίσιο. Και το τρίτο θεσμικό όργανο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα δούμε λοιπόν και την απόφαση για το θέμα αυτό, να δούμε τι, ποιος θα εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν ε, ήθελα να σας πω ως ανακοινώσεις Προέδρου. Ο Τζόρτζ και οι Μερσέντες ε, θέλουν το λόγο. Τζόρτζ. Μία ερώτηση έχω κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Στι διαπραγματεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit έχω την αίσθηση ότι η Ιρλανδική Δημοκρατία έχει σκληρύνει τη θέση της. Έχετε κι εσείς αντίστοιχη άποψη. Δεν ξέρω εάν μπορώ να πω έτσι ομά ναι, αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ, αλλά αυτό ακούγεται. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει, αλλά έχω ακούσει κι εγώ αυτή την άποψη δεν ε, φάνηκε κάτι τέτοιο στις συζήτηση της Κόζακ ή Mercedes Μπρέσο. Για το πρώτο σημείο, για το χρόνο της ψηφοφορία δεν έχει σχέση με τις ανακοινώσεις σας. Ήθελα απλώς ε, να ζητήσω ονομαστική κλίση για το ψήφισμα. Νόμιζα ότι είχατε τελειώσει, γι' αυτό ε, ζήτησα το λόγο. Είναι για το επόμενο σημείο. Ωραία. Έχουμε μια πρόταση της ομάδας σας να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για τις προφορικές ερωτήσεις που αφορούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος σε αυτή την πρόταση. Δεν βλέπω κάποιον. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε όπως ζητά η ομάδα των σοσιαλιστών. Είναι σύνομο με τον κανονισμό, επομένως μπορούμε να κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. To test the machine. Να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. Μια δοκιμή πρώτα. Αν έχετε την καλοσύνη, να τοποθετήσετε τις κάρτες σας στη συσκευή. your Δεν δοκιμάσατε όλη την κάρτα σας, αλλά νομίζω μεγάλοι άνθρωποι είστε, ξέρετε τι κάνετε. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ρωμάν Χαουρέκη, ο, ο Ραμόν δεν είναι παρόν. Να θυμίσω μόνο, ε, επειδή δεν μπορεί εκείνος να πάρει το λόγο, να σας θυμίσω ότι είναι ένα θέμα που συζητιέται από τον ε, Μάρτιο 2014, από την ε, τελευταία ολομέλεια της προηγούμενης θητείας. Δεν υπήρχε βούληση από πλευράς του Συμβουλίου. Τελικά η Σλοβακική Προεδρία είχε μια εξαιρετική ιδέα. Οι νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων ε, διαπραγματεύτηκαν επί αρκετές, ε, αρκετούς μήνες. Ε, τελικά καταλήξαν σε μια καλή πρόταση και ε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Η προφορική ερώτηση, λοιπόν, σχετίζεται με αυτήν την ιδέα να κινητοποιηθούν τα δύο θεσμικά όργανα. Έχουμε λοιπόν δύο ψηφοφορίες. Ψηφοφορία για το σχέδιο προφορικής ερώτησης με συζήτηση προς το Συμβούλιο. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ε, περισσεύει μια ψήφος του ΕΛΚ. Μου λένε. Δύο ψηφοφορίες έχουμε λοιπόν. Δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά πάντως έχουμε μία ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚ από ό,τι θα έπρεπε. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Λήξη της ψηφοφορίας. Η 21 ψήφοι υπέρ, μια αποχή. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Ε, και ψηφοφορία πάνω στη δεύτερη ερώτηση. Έναξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιος απέχει λοιπόν. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία και προχωράμε σε ένα θέμα που είχαμε προγραμματίσει για τις 10 και 4. Χρειαζόμαστε παρουσία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συνάδελφοι ελπίζω να είναι εδώ. Αλλιώς μάλλον πρέπει να περιμένουμε λίγο. Yes, they, it's her,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 στις παρουσιάσεις. Ε, Βάρβαρα, μήπως ε, θέλεις όμως να κάνεις πρώτα μια εισαγωγή. Δεν ε, βλέπω που είναι. Μιλάει. Θα ήθελες να κάνεις μια εισαγωγή ή να δώσω κατευθείαν το λόγο στους ομιλητές μας. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας τους προσκεκλημένους της Βαρβάρες ή μάλλον της Επιτροπής. Ε, θα μας παρουσιάσουν ε, ε, την υλοποίηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε εδώ μαζί μας τον καθηγητή Ολιβιέ Σχούτερ. Σε παρένθεση μου έχουν γράψει εδώ πώς προφέρεται το όνομα. Καλό λοιπόν τον καθηγητή Ολιβιέρ Σκούτερ, Σούτερ διορθώνει η πρόεδρος. Πάσε πτώση, ξέρετε ότι για σας μιλάμε. Βλέπετε σε ένα τέτοιο πολιτισμικό περιβάλλον, ε, συχνά μας δυσκολεύουν τα ονόματα. Λοιπόν, είσαστε ο πρώτος ε, ομιλητής και παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη μας πείτε και πώς προφέρετε το όνομά σας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ε, η συζήτηση να οδηγήσει σε εξίσου ε, έντονες συζητήσεις με αυτήν που προκαλεί η προφορά του ονοματός μου. Ε, λέγομαι λοιπόν ε, Ολιβιέρ Σούτερ και... Η έκθεση που παρουσιάζεται για να υποστηρίξει την έκθεση της κυρίας Πινέλη για τον χάρτη των θεμελιωτών δικαιωμάτων, στόχο έχει να δείξει πώς μπορεί ο χάρτης των θεμελιωτών δικαιωμάτων να επηρεάσει την νομοθεσία και τη διαμόρφωση πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους τομείς. Η μελέτη αυτή είναι αρκετά εκτενής, έξι τομείς καλύπτει. τους οποίους ε, προφανώς δεν θα μπορέσω να σας παρουσιάσω αναλυτικά κατά αυτήν την ε, εισαγωγική παρουσίαση. Εξετάζει η μελέτη πώς λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων με μελέτες αντικτύπου. και τη φροντίδα από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να φροντίσει να μην ε, παραβιάζουν το χάρτη μελιωτών δικαιωμάτων ε, οι νομοθετικέ της προτάσεις. Βλέπουμε πώς μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική διακυβέρνηση, <clears throat> πώς επηρεάζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς εφαρμόζονται τα μέτρα από τα κράτη-μέλη τι ρόλο παίζει στις εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τι ρόλο παίζει όσον αφορά ε, τα ένομα μέσα προσφυγής. Αποφάσισα λοιπόν να επικεντρώσω τη μελέτη μου σε τρία από αυτά τα θέματα και θα ξεκινήσω από την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έναν τομέα χωρίς δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συστηματική αναγνώριση ε, του ότι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να παίξει ρόλο η οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ξεκινάει κάτι τέτοιο και το δικαστήριο τονίζει την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να λάβουν υπόψη τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει όμως συστηματική πρακτική μέχρι τώρα. Η κοινωνικο-οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύπλοκο θέμα. Γι' αυτό είναι δύσκολο για μη ειδικού να συμμετέχουν στη συζήτηση, αλλά μπορούμε εύκολα να τη συνοψίσουμε. Υπάρχουν τέσσερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρακολουθεί τα κράτη-μέλη και να διασφαλίζει την οικονομική σύγκληση, ιδιαίτερα εντός της Ευρωζώνης. Καταρχάς, λοιπόν, έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεύτερον, έχουμε τους ειδικού κανόνες που ισχύουν για κανόνες που λαμβάνουν η οικονομική υποστήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό 472 κάθετος 2013. Τρίτον, από το, την 1η Μαΐου 2012 έχουμε την συνθήκη για την σταθερότητα, των συντονισμό και την διακυβέρνηση εντός της ΟΝΕ που επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη-μέλη και τέλος έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, Σταθεροποίησης. Ένα ε, δούνου του για την Ευρωζώνη. Η μελέτη προσπαθεί να εξετάσει πόσο ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων επηρεάζει την χρήση αυτών των εργαλείων. Και υπάρχουν πολύ σημαντικά επιχειρήματα ώστε ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων να παίξει πιο σημαντικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική διακυβέρνηση. Καταρχάς ε, το δικαστήριο στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016 ε, εξόδωσε απόφαση ε, στην υπόθεση Ledra Advertising που είχε να κάνει με τη διάσωση της Κύπρου και συμπεριελάμβανε το λεγόμενο κούρεμα Ε, καταθέσεων Κυπριωτών. Και αυτοί προσέφηγαν στο δικαστήριο διότι είπαν ότι ε, έχει προσληθεί το δικαίωμα ε, της ιδιοκτησίας τους και το δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον χάρτη ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, το ίδιο είπε και ο Γενικό Εισαγγελέα. Δεν ε, προχώρησε τόσο όμω ώστε να πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλλει σε άλλου, δηλαδή στην Κύπρο, ε, να συμμορφώνεται με τον χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων, αλλά αυτή είναι η ουσία της ε, απόφασης αυτής, ότι ε, η απόφαση αυτή απευθύνεται στα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπόψη και εκτός των θεσμικών οργάνων, για παράδειγμα ε, στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ε, και θα πρέπει ακόμα και εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να λαμβάνεται υπόψη αυτό, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Υπάρχουν επίση ισχυρά οικονομικά επιχειρήματα για την ενίσχυση του ρόλου του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τομέα αυτών. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στην διάσκεψη κορυφή του Γκέτεμπορκ ε, υιοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ένα από του βασικού λόγου που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθετήθηκε τελικά ήταν ότι τα δικαιώματα αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο ε, σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και μπορούν να βοηθήσουν ε, στην ε, διασφάλιση σταθερότητας κατά την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πράγματι πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την παρουσίαση του πυλώνα τόνισε τον ρόλο των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην προσέλκυση επενδύσεων ε, στην διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Και γι' αυτό υπάρχουν και οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου των κοινωνικών δικαιωμάτων ε, στην οικονομική διακυβέρνηση. Η μελέτη μας κάνει κάποιες συστάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να λαμβάνεται υπόψη καλύτερα ο πυλώνας ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Και ε, υιοθετούνται συστάσεις αναχώρα κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί κάθε χρόνο τις συστάσεις της στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης ε, που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διατακτικά στοιχεία του χάρτη. Ε, υπάρχει ήδη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχει συνείδηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο. Μέχρι σήμερα όμως ε, δεν υπάρχει ε, ρητή αναφορά του αντίκτυπου σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και κάτι τέτοιο μπορεί να καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της κατά διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεύτερον, όσον αφορά το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ε, αναφέρομαι στη συνθήκη του 2012 για την ε, διακυβέρνηση. Τα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό εποπτεία δεν επιτρέπεται να έχουν ε, έλλειμμα παραπάνω από ε, μια συγκεκριμένη τιμή, μπορούν όμως να αποκλίνουν από την πορεία που έχουν ανακοινώσει σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων. Άρθρο 3, 3β της ε, συνθήκης. Αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις ορίζονται με αρκετά περιοριστικό τρόπο στο πλαίσιο του άρθρου 3.3β. Μας, η μελέτη μας συστήνει αυτή, αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις να συμπεριλαμβάνουν και τη δυνατότητα την ανικανότητα ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί χωρίς να παραβιάζει τις υποχρεώσεις ε, σύμφωνα με τις ε, κοινωνικές διατάξεις του χάρτη. Πρόκειται λοιπόν για εξαιρετικέ περιστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν αλλάξει την πορεία που έχει ανακοινώσει, μπορεί να χρειαστεί να μειώσει συντάξει, να περιορίσει τα, τις γιατρικές παροχές κλπ. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι κοινωνικές περιστάσεις να λαμβάνονται υπόψη ε, όταν ένα κράτος μέλος ε, ζητάει να αποκλίνει από τον, την πορεία που έχει ανακοινώσει. Τρίτον, ε, σε περίπτωση που ο κράτος μέλος βρίσκεται υπό εποπτεία επειδή έχει λάβει ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ε, παραμείνει βιώσιμο το χρέος. Το μνημόνιο που διαπραγματεύονται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό το απέτησε το ε, δικαστήριο σε αυτήν την απόφαση της Lidra Advertising στην οποία ήδη αναφέρθηκα και μάλιστα στην υπόθεση Φλωρέσκου της 13ης ε, Ιουνίου του 2017 που εξορισμού δεν, συμπεριλα... Ε, δεν τη συμπεριλάβαμε στην ε, μελέτη μας, αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με το Μνημόνιο Ρουμανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το ε, μεγάλο περιθώριο που δόθηκε στην Ρουμανία ε, θεωρήθηκε ότι ε, η Ρουμανία ενεργεί στα πλαίσια της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαμόρφωση των συντάξεων και αυτό θα πρέπει να, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να παραβιάζει τα κοινωνικά δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να, να ενισχυθεί στο μέλλον. Γι' αυτό ε, εκπονούμε αυτή τη στιγμή κατευθυντήριες αρχές ε, που θα εκπονηθούν από τον ε, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζουμε, ο χάρτης θεμελιωτών δικαιωμάτων ε, ισχύει όχι μόνο για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισχύει και για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρακτική όμως εντός των οργανισμών ε, διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς οι διάφοροι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εφαρμόζουν ή όχι τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και προσπαθούμε να επισημάνουμε κάποιες καλές πρακτικές που προέκυψαν από τη σύγκριση αυτή. Ε, και προτείνουμε εδώ έξι βασικούς κανόνες και το ονομάζω six-pack με πολύ προκλητικό τρόπο ε, διότι αναφέρεται στο πώς μπορούν τα κράτη τα, οι οργανισμοί να λάβουν υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα στη δουλειά τους. Για παράδειγμα, ε, ο πρώην Frontex, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και η ΕΑΣΟ Είναι ενδιαφέρον πόσο διαφορετικά προσεγγίζουν τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επικροτούν τον χάρτη για να ενισχύσουν τον ρόλο τους. Έξι λοιπόν είναι αυτές οι καλές πρακτικές. Ε, οι οργανισμοί αυτοί λοιπόν μπορούν να υιοθετήσουν στρατηγική θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως έχει ήδη γίνει από την Frontex όπως περιγράφουμε στη μελέτη μας. Δεύτερον, θα μπορούσαν ή θα έπρεπε μάλλον ε, να αναφέρουν ε, τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στον κώδικα δεοντολογίας τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς που να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων εντοπίζεται αμέσως και εξετάζεται θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένας ε, αξιωματούχο θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, που να ενεργεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο προσωπικό και ε, να παρακολουθεί εντός του οργανισμού περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν. Πέμπτον, καλή πρακτική είναι να υπάρχει συνεχής διάλογος με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς πάνω σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προφανώς γίνεται και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά όπως γίνεται και από άλλους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένης της Frontex. Έκτον, στο βαθμό που οι οργανισμοί αυτοί συχνά ε, συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να αναφέρονται να συμπεριλαμβάνονται στους όρους αναφοράς ε, του διαλόγου με αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες στα μνημόνια που συνάπτονται με εθνικές διοικήσεις. Αυτές λοιπόν είναι έξι συστάσεις που προκύπτουν από την εξέταση του πώς οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ε, ενσωματώνουν στη δουλειά τους ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης ε, θα ήθελα να επιστήσω την ε, προσοχή της Επιτροπής σας σε, ένα ακόμα θέμα. Ε, την πρόσβαση σε ένομα μέσα, σε ένδικα μέσα και όπως θα γνωρίζετε, όταν διαπραγματευτήκαμε την, τη συνθήκη, Η πρόσβαση σε ένδικα μέσα τροποποιήθηκε στο άρθρο 263 παράγραφος 4, το πρώην δηλαδή άρθρο 230 της ε, συνθήκης. Τροποποιήθηκε ώστε να διασφαλίζεται ότι όποιος επηρεάζεται άμεσα από ε, κανονιστική πράξη των ε, θεσμικών οργάνων θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει ακύρωση της πράξης μεταξύ άλλων για να διασφαλίσει τη μη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το πρόβλημα ήταν ε, ότι αυτό ήταν λάθος ε, στην ε, σύνταξη της συνθήκης της Λισαβόνας, διότι δεν αναφέρονται ρυθμιστικές πράξεις το 2003 και Γι' αυτό περιέργως έχουμε εδώ αναφορά σε κανονιστικές πράξεις χωρίς να υπάρχει ο σχετικός ορισμός στις συνθήκες. Ωστόσο, το δικαστήριο έχει ερμηνεύσει με περιοριστικό τρόπο ε, αυτό το θέμα στην απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2013 Ινουίτ, Ταπιρίτ, Κανατάμι και άλλοι. Λέει λοιπόν ότι ενώ άτομα που επηρεάζονται από μία πράξη μπορούν να αρτήσουν ακύρωση της πράξης στο δικαστήριο, αυτό δεν ισχύει για νομοθετικές πράξεις. Δηλαδή νομοθετικές πράξεις που έχουν υιοθετηθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης, όπου συνομοθετούν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Αυτό όμως ε, οδηγεί σε νομικό κενό, διότι όταν ε, υιοθετείται μια νομική πράξη, αυτό που επηρεάζει κάποια άτομα, τα άτομα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στο δικαστήριο για να ζητήσουν την ακύρωση μιας τέτοιας νομοθετικής πράξης. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε το ε, κενό αυτό. Στη μελέτη ισχυριζόμαστε ότι όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει να κλείσει από τα κράτη-μέλη που έχουν υποχρέωση ε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, και σύμφωνα με το άρθρο 19 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν ένδικα μέσα επαρκή ώστε να διασφαλίζεται πραγματική νομική προστασία στους τομείς που καλύπτονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό είναι υποχρέωση των κρατών μελών να οργανώσουν ε, τις αρμοδιότητες των ε, εθνικών τους δικαστηρίων, τη δικαιοδοσία τους έτσι ώστε να επιτρέπουν ε, προσφυγές στα δικαστήρια ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική νομική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη θα πρέπει να επιτρέπουν σε άτομα να ζητούν νομική προστασία ακόμα και πριν εφαρμοστεί κάποιο μέτρο που να τους επιβάλλει κάποια κύρωση, για παράδειγμα, και δεν θα πρέπει να ε, πρέπει πρώτα να παραβιάσουν τον νόμο για να, τον, ε, για να προσφύγουν κατά του στο δικαστήριο. Από τη στιγμή δηλαδή που εφαρμόζεται ε, ένας νόμος και οδηγεί σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει κανείς από το δικαστήριο έγκυρη ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να επιτρέψει στο δικαστήριο να αποφασίσει αν η νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ή αν πρέπει να ακυρωθεί. Έχουν εξεταστεί οι τρόποι πρόσβασης ε, στα δικαστήρια των κρατών μελών Ε, στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχει ένα ακόμα κενό στο σύστημα ένδικων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχει να κάνει με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, την ΚΕΠΑ. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου είναι περιορισμένη στον τομέα αυτόν. Αυτό σκόπιμα έγινε με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, διότι υπήρχε η γνώμη ότι το δικαστήριο δεν θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί πολύ στενά ε, τους τομείς ε, εξωτερικών σχέσεων. Αλλά κάποιες φορές υπάρχουν επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ που μπορεί να επηρεάσουν τα, ε, ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα ατόμων. και υπάρχει το άρθρο 275 της ε, Συνθήκης ε, για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπου περιγράφονται κάποια περιοριστικά μέτρα, κυρώσεις δηλαδή κατά τρομοκρατών ή υπόπτων για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγή στο δικαστήριο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι μπορεί να χρειαστεί να λογοδοτήσουν σε δικαστήριο, μπορεί να ε, θέλουν να ε, εκδώσουν κάποια δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη, αλλά εξαιρείται ε, από, τον έλεγχο και τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ μπορεί να δεχτούν προσφυγή στο δικαστήριο. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια σημαντικά σημεία από την ε, μελέτη αυτή που στόχο έχει να βοηθήσει την κυρία Σπινέλη στην εκπόνηση της εκθεσή της και προσλέπω στην συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση, θα ήθελα να μου δώσετε μια διευκρίνηση. Δεν μιλήσατε για ε, άτυπες ομάδες όπως το Eurogroup για παράδειγμα. Πώς τους κατατάσσετε. Θεωρείτε πως είναι φορέας, υπηρεσία ή ε, ουσιαστικά ε, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση σεβασμού της χάρτας. Το Eurogroup δεν αποτελεί επίσημο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα μέτρα τα οποία εγκρίνονται από το Eurogroup και οι αποφάσεις που λαμβάνει, όντως περνάνε ως μέτρα από τα κράτη-μέλη στα οποία απευθύνεται το Eurogroup. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά όντως εμπίπτουν ε, στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομίζω ότι αυτό απορρέει από την απόφαση Φορέσκου ε, και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον υπονοείται από άλλες αποφάσεις επίσης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμία ε, αμφιβολία πως θα πρέπει το Γιώργο να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του σεβασμού της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, παρόλο που το ίδιο δεν αποτελεί κάποιο θεσμικό όργανο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 51. Σας ευχαριστώ πολύ. Περάσουμε λοιπόν την κυρία εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα μας δώσει τη δική της άποψη για το θέμα αυτό. Ξέρω πως θα μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία που έχετε αποκομίσει από το Συμβούλιο για το σχετικό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότυπα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και επίσης θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να ε, ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Σούτερ για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, όπως είπατε μάλλον εσείς, αυτή τη στιγμή έχω την ε, προεδρία της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και για τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα εργασία η δική μα είναι υπεύθυνη για την εργασία προετοιμασία κατά την νομοθετική ε, προσπάθεια που κάνει το Συμβούλιο στον χώρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των πολιτών και ελεύθερη κυκλοφορία, όπω επίση και για όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την προώθηση και συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα με καλέσατε να πάρω το λόγο για δύο κυρίως θέματα. Πρώτα απ' όλα για τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μεθοδολογικά βήματα που θα λάβουμε για να ελέγξουμε τη συμβατότητα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στα βήματα προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το δεύτερο θέμα είναι η συνεργασία στο Συμβούλιο όποτε ε, προκύπτει θέμα με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το θέμα λοιπόν της σημερινής συζήτησης έχει να κάνει με την εφαρμογή ε, της χάρτας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτής. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να μιλήσω εντάχει και για την εφαρμογή της χάρτας σε αυτό το δεύτερο εξάμεινο της ε, φετινής χρονιάς. Και το τι, έχουμε, το τι έχουμε κάνει στην ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο γύρω στο Μάη δημοσιεύει μια έκθεση για την πορεία της ε, εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η σχετική υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα επίσης μια φορά το χρόνο εκδίδει μια έκθεση όπου περιγράφει τις βασικές εξελίξεις σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασιζόμενοι σε αυτή αυτές τις δύο εκθέσεις κάθε χρόνο το Συμβούλιο εγκρίνει ε, συμπεράσματα για το πώς εφαρμόζεται η χάρτα. Η μέχρι τούδε διαδικασία της έγκρισης των συμπερασμάτων το πρώτο εξάμεινο της χρονιάς συνήθως δεν είχε προσφέρει την βέλτιστη ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση εξαντλητική για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά φέτος η συζήτηση και η έγκριση των συμπερασμάτων αναβλήθηκε και θα λάβει χώρα τώρα το δεύτερο εξάμεινο. Άρα λοιπόν ακόμα βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η παρουσίαση των εκθέσεων και η συζήτηση που θα γίνει ε, αυτών στην ομάδα εργασίας μας οδήγησε στο εξής συμπέρασμα. Καταρχήν, είναι ένα θέμα που ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη, γίνεται πάρα πολύ ζωντανός διάλογος. Στη συνάντησή μας του Οκτωβρίου στο Συμβούλιο κάναμε μια πολιτική συζήτηση για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εδώ θα συμπεριλάβω μια ανταλλαγή απόψεων που σημειώθηκε με τον Διευθυντή ε, της Υπηρεσίας για τα θεμπελιώδη Δικαιώματα, τον κύριο Μάικλ Φλόρετσι, ο και μετά από τη συζήτηση αυτή εγκρίναμε και τα συμπεράσματα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδικών Δικαιωμάτων κατά το έτος 2016. Τα συμπεράσματα αυτά αποδεικνύουν πως χρειάζεται να ενσωματώσουμε απολύτως τα θεμελιώδη δικαιώματα στην αξιολόγηση και προετοιμασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα συμπεράσματα μας υπενθυμίζουν δε πως οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα μεθοδολογικά βήματα που θα εφαρμοστούν έτσι ώστε να εξεταστεί η συμβατότητα των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ε, τις όσες κάνουν τα ε, όργανα προετοιμασίας νομοθεσίας του Συμβουλίου ε, είναι μια ε, διαδικασία η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές χρησιμεύουν γιατί στο Συμβούλιο έχουμε πάνω από 150 ομάδες εργασίας που ασχολούνται με πολύ διαφορετικά αλλά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Άρα λοιπόν οι διάφοροι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες εργασίας ενδεχομένως δεν έχουν ε, φυσική εμπειρία για να μπορούν να ελέγξουν τη συμβατότητα των όσων ε, εργασιών κάνουν και το πώς αυτά ε, σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα λοιπόν αυτά τα όργανα του Συμβουλίου θα πρέπει, το λένε και τα συμπεράσματα, να εξετάσουν με πολύ σοβαρότητα οποιαδήποτε παρέμβαση στις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Και γι' αυτό τον πολύ πρακτικό λόγο είναι σημαντικό οι προτάσεις που γίνονται να συμμορφώνονται με την χάρτα γιατί ε, διαφορετικά ε, ε, θα τα καταρρύψει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης, στόχος μας είναι να ευαισθητοποιηθεί το Συμβούλιο και ομάδες εργασίας αυτού για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για να προωθήσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, η γραμματεία του Συμβουλίου τα συμπεριλαμβάνει, συμπεριλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές στις γενικές εκπαιδεύσεις που κάνει σε κάθε καινούργιο καινούργια Προεδρία του Συμβουλίου που αναλαμβάνει καθήκοντα και επίσης στην αρχή κάθε Προεδρίας η Προεδρία καλεί ε, της ε, προεδρίες όλων των υπολείπων ομάδων εργασίας να ε, μοιράσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές σε όλους τους υπεργνώμονες. Επίσης, η σχετική υπηρεσία προσφέρει ε, επιμορφωτικές ε, ημερίδες στα κράτη-μέλη, στις αντιπροσωπείες αυτών και σε όλο το προσωπικό και οι κατευθυντηρίες γραμμές δίνουν ακριβώς μια κατεύθυνση για την όλη διαδικασία ε, εξέταση, συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το fundamental rights checklist ε, tool to facilitate the assessment. Και υπάρχει και ένα σχετικό ερωτηματολόγιο checklist, μια κατάσταση ελέγχου, έτσι ώστε κάθε πρόταση να μπορεί να εξεταστεί σε συνάρτηση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση. Επίσης, το checklist αυτό μπορεί κανείς να εντοπίσει αν υπάρχει συσχετισμός με θεμελιώδη δικαιώματα και πώς μπορεί κανείς να εξετάσει κατά πόσο μια πρόταση ευθυγραμμίζεται με ε, τη χάρτα ή όχι. Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν κάποιες εξηγήσει, δίνουν κάποιο ε, υλικό που βασίζεται στην ομολογία και δίνουν και κάποιες οδηγίες για το πώς θα πρέπει ε, κανείς να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Έχουμε την Charterpedia, την οποία προετοίμασε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, σε συνεργασία με την υπηρεσία, σχετική υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπου έχουμε διάφορες πρακτικές, νομολογίες, αποφάσεις κτλ, πρακτικές συμβουλές που σχετίζονται με τη χάρτα. Η ομάδα εργασίας δεν μπορεί να προσφέρει στις άλλες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου νομική αρρωγή για το πώς θα εντοπίσουν και θα ενσωματώσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά υπάρχει νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, η οποία γνωμοδοτεί ε, για νομικά θέματα και προσφέρει νομική συνδρομή και αναλαμβάνει το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά εμείς ενημερώνουμε έτσι ώστε να γίνει κάποια συζήτηση, να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν σε άλλες ομάδες εργασίας έτσι ώστε να είναι όλοι ενήμεροι. Και αυτό βέβαια γίνεται και αντίστροφα έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, εμπλέκεται στην ε, νομοθετική διαδικασία, βεβαίως με συμβουλευτικό ρόλο. Και πολύ συχνά η υπηρεσία αυτή προσκαλείται το Συμβούλιο έτσι ώστε να ενημερώνει και τους εμπειρογνώμονες αλλά και τους υπουργού για θέματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα για τη συνεργασία. Η Προεδρία της Εστονίας και το πώς συνεργαστήκαμε με την Υπηρεσία Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Να σας πω πολύ συγκεκριμένα πώς έχουμε παραδείγματα τα οποία μπορώ εδώ να σας παρουσιάσω. Όπως όλες οι προεδρίες, έτσι και εμείς, συμφωνήσαμε τη συνεργασία μας με την υπηρεσία πολύ πριν ξεκινήσει η προεδρία μας με ποιο τρόπο. Η υπηρεσία μας επισκέφθηκε στη χώρα μας, συζητήσαμε τη δυνατότητα συνεργασίας και η υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να σας πω πως κάνει κάτι αντίστοιχο με κάθε προεδρία που ξεκινάει. Το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει καταθέσει ε, επεξηγηματικά σημειώματα και ε, βοήθεια για θέματα τα οποία τρέχουν στα πλαίσια του διαλόγου για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο για τα μίντια, για τον πλουραλισμό, ε, για τα όσα μπορούν να ισχύσουν αυτό το χώρο στην ψηφιακή και να σας πω πως η υπηρεσία κατέθεσε και μία παρουσίαση στην, στο σεμινάριο εμπειρογνωμόνων που κάναμε το Ιούλιο στις Βρυξέλλες και επιπλέον έγινε και μία θεματική συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με μια ανταλλαγή απόψεων με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και πρέπει να σας πω πως η υπηρεσία αυτή μέσω του Διευθυντή της συμμετείχε στην εισαγωγική ε, ανταλλαγή απόψεων, στην ε, συζήτηση πολιτικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα που έγινε κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου του Συμβουλίου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Επίσης να σας πω πως στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, σε σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπηρεσία κατέθεσε ε, μία έκθεση για την εξωτερική και εσωτερική συνοχή της πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Να σας πω πως στα φετινά συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εφαρμογή της χάρτας η υπηρεσία λέει πως το Συμβούλιο αναγνωρίζει το ρόλο ε, της ε, σχετικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα όσα έχει στο καταστατικό της και δέχεται τις συμβουλές της όπως επίσης και την πραγματογνωμοσύνη της ε, για τα θέματα αυτά και το κάνει ήδη εδώ και μια δεκαετία. Επίσης θα πρέπει ε, η υπηρεσία να ενισχυθεί ε, στο ρόλο της αυτό μέσω συνεργειών και συνεργασίας μέσω δικτύων επαφών, σημείων επαφών με κυβερνητικές εργανώσεις, με την κοινωνία των πολιτών ε, και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων για τη βέλτιστη εφαρμογή της χάρτας και την κοινοποίηση ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων προς το ευρύτερο κενό. Τέλος, η υπηρεσία αυτή αποτελεί ε, και το think tank του Συμβουλίου για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και προσφέρει στα κράτη-μέλη μια καλή πηγή ε, πραγματογνωμοσύνης ε, και ενημέρωσης. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τουπάη και τώρα έχουμε ένα συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διάθεση ε, Jazz, τη Λίντα Μαρία Ράβου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Επιτροπή ΑΦΚΟ που μας προσκάλεσε εδώ σήμερα για να μοιραστούμε την εμπειρία μας και να σας ε, πούμε την άποψή μας και να ακούσουμε την ε, τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εφαρμογή της χάρτας ε, σε θεσμικό πλαίσιο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ολιβιέντε Ντεσούτερ για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και την παρουσίασή του σήμερα. Οι παρατηρήσεις του όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και ε, τα θέματα που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητες ε, που ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλά και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό πολιτών και τη συνέχεια που δίνεται στις αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδίω στην απόφαση Λίδρα, είναι πάρα πολύ σημαντικές και νομίζω ότι αυτά έχουν μεγάλη σημασία και για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που όπως ξέρετε είναι πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σημαντικές και οι παρατηρήσεις όσον αφορά το ρόλο και τις ευθύνες των ευρωπαϊκών ε, οργανισμών και υπηρεσιών Ιδίως σε μια στιγμή που υπάρχουν κάποιοι πολύ σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και υπηρεσίες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που την χάνουν σε αυτή τη στιγμή. Ο νέος οργανισμός που αντικαθιστά το Frontex για παράδειγμα ε, και ο νέος ρόλος και η νέα εντολή για τις νέες του δραστηριότητες αλλά και ο ΕΑΣΟ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου, ε, το ΙΓΙΟΛΙΣΑ και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Είμαι βέβαιος, βέ, βέβαιη ότι τα όσα συζητάτε θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα άλλα θεσμικά όργανα και τους ίδιους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες. Και επίσης ε, διαπιστώνουμε ότι ο Οργανισμός Θεμελιδιών Δικαιωμάτων διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και παρέχει καθοδήγηση και εκπαίδευση σε κάποιους ε, ε, βασικού εταίρου στον τομέα των ιστορικών υποθέσεων, όπω για παράδειγμα το Frontex. Και είμαι βέβαιη ότι αυτό θα συνεχιστεί και αυτή είναι μια πολύ σημαντική ε, διαδικασία την οποία υποστηρίζουμε. Όσον αφορά τη δική μου την παρουσίαση, σήμερα μου ζητήσατε να πω δύο λόγια για τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εξασφάλιση εφαρμογής της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την εμπειρία μας, τις πρακτικές μας και θα πω και δύο λόγια για κάποια επιτεύγματά μας, αλλά και προκλήσεις ε, στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πολύ καλά επεσήμανε η μελέτη του κυρίου Ντεσούτερ, έχει αρκετά εργαλεία για να ε, διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται ε, οριζόντια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στα θεσμικά όργανα και ε, σταδιακά έχουμε βελτιώσει και τη μεθοδολογία μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όντως εφαρμόζεται στην πράξη ο χάρτης σε ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έλεγα ότι το πλαίσιο και αυτά τα εργαλεία και αυτή τη στρατηγική είναι ε, μια στρατηγική η οποία αποκαλείται στρατηγική των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο εγκρίναμε το 2010 για την αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο στόχος ήταν καταρχάς να ανταποκριθούμε στις νέες αξίες ε, που προσλαμβάνει ο χάρτη με τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα το 2009 και να δώσουμε και κάποιε κατευθυντήριες γραμμές ώστε αυτέ οι νέες ε, δεσμευτικές ε, ε, πτυχές που αποκτά ο χάρτης θα μπορέσουν να έχουν και κάποιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει τα καθήκοντά της και τις ευθύνες της. Θέλαμε λοιπόν καταρχάς να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση και προώθηση του χάρτη στην νομοθετική ε, διαδικασία, να εγγυηθούμε δηλαδή ότι ε, λαμβάνονται τα κατάλληλα ε, βήματα ώστε να συμπεριλαμβάνεται και να λαμβάνεται υπόψη ο χάρτη σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας και την άσκηση της εξουσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει νομοθετικές πράξεις να εξασφαλίσουμε το σεβασμό του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά επίσης και να παρέχουμε πληροφορίες προς το ευρύ κοινό και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πεδίο εφαρμογής του χάρτη και για την προστασία που παρέχει, καθώς επίσης και πληροφορίες ε, για ε, διαθέσιμα ε, μέτρα, αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό φυσικά ε, για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο στην εφαρμογή του χάρτη κάθε χρόνο, ε, το οποίο γίνεται μεταξύ άλλων και μέσω της δημοσίευσης μιας ετήσιας έκθεσης την οποία ανέφερε και η συνάδελφος από το Συμβούλιο ήδη. Πολύ σύντομα, διότι είμαι βέβαιη ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πώς έχει διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι και αντίστοιχη με αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος από το Συμβούλιο όσον αφορά τον κατάλογο ελέγχου των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και να σας πω απλώς ότι επί τη βάση αυτής της στρατηγικής και του χάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κάποιες πρακτικές ε, ε, οδηγίες για το πώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης της αξιολογής επιπτώσεων. Αυτό δημοσιεύτηκε το 2011 και στόχο έχει να εξασφαλίσει ότι ο χάρτης των θερμολογιδών δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη σε όλη την νομοθετική διαδικασία ακόμα και πριν γίνουν οι αξιολογίες των επιπτώσεων ε, στα προκαταρκτικά στάδια της προετοιμασίας μιας νομοθεσίας ε, και στις προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις ε, και στις ίδιες εκτιμήσεις των επιπτώσεων και από εκεί και πέρα στη σύνταξη και κατάρτιση των προτάσεων και στη διαπραγματευσή τους. Ενισχύσει και δε περαιτέρω ο μηχανισμός αυτός από τη δέσμη μέτρων για την καλύτερη νομοθεσία του 2015 και τη δέσμη μέτρων του 2017 για την καλύτερη νομοθεσία και μάλιστα τώρα συνοψίζεται σε μία εργαλειοθήκη, την υπαριθμών 28, η οποία παρέχει ουσιαστικά ένα εύχριστο οδηγό ε, των όσων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα θεμελιώδη δικαιώματα για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και ε, συμπληρώνει αυτές τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές ε, οι οποίες εξετάζουν όλα τα θέματα με λίγο πιο διεξοδικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή βεβαίως εφαρμόζεται σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και παράλληλες προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αντίκτυπο ε, για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και όσων διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, κάποιες πράξεις οι οποίες ε, έχουν κάποια επιρροή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργαλειοθήκη λοιπόν αναφέρει και τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εγκρίθηκαν πέρσι για την υποχρέωση εξορθολογισμού και συμπερίληψης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εμπόριο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική και οι επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο ε, αποτελούν ένα σύστημα ε, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης ε, με τρεις πτυχές αν θέλετε, τρεις διακλαδώσεις, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, να μην λαμβάνονται δηλαδή μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να παρέμβουν ε, χωρίς λόγο ε, στο όσα προβλέπει ο χάρτης. Όπως είπα από την αρχή, λαμβάνονται υπόψη όλα από την ε, εκτίμηση επιστε... επιπτώσεων μέχρι την κατάρτιση της νομοθεσίας και τη διαπραγμάτευση, αλλά επίσης να προωθούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω τη χρήση τη εξουσίας ε, υποβολής προτάσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορου τομεί ε, οι οποίοι ε, μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία και το υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για παράδειγμα τον τομέα της έλλειψης διακρίσεων, της προστασίας δεδομένων, της ποινική δικαιοσύνης και κυρίως τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορημόνων. Ε, αλλά υπάρχει και μια τρίτη πτυχή που είναι αυτή της προστασίας του ίδιου του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή να εξασφαλίζουμε ότι εφαρμόζεται ιδίως ε, ε, όσον αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον πράξεων των κρατών μελών. Και φυσικά ε, λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο χάρτη και επίσης και εδώ χρησιμοποιώ κάτι το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον στην ε, έκθεση του καθηγητή De ε, και άλλα πηγέ ε, άλλες πηγές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλα εργαλεία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμφαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άλλα διεθνή μέσα αλλά φυσικά και τα συντάγματα των κρατών μελών από τα οποία μεταξύ άλλων έχουμε εμπνευστεί και το χάρτη των θεμελωδών δικαιωμάτων. Και το λέω αυτό βεβαίως διότι αποτελεί υποχρέωση και από τα ίδια τα δικαιώματα του χάρτη. Στις γενικές διατάξεις του χάρτη και κυρίως τα άρθρα 52 και 53 και μάλιστα και στις αιτιολογικές ε, σκέψεις που αφορούν τις συγκεκριμένες διατάξεις του χάρτη, είναι σαφές ότι όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη δεδομένου ότι δεσμεύονται από το χάρτη, πρέπει να τον εφαρμόζουν και ε, βάσει ε, διεθνών ε, και άλλων μέσων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δύο λόγια όσον αφορά τις λεγόμενες πτυχές προστασίας, δηλαδή την ε, εφαρμογή των υποχρεώσεων των κρατών μελών ε, να λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης ε, Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει διαδικασίε επί όταν παραβιάζεται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τα κράτη-μέλη. Αυτό περιλαμβάνει και τι διατάξει του χάρτη, όταν η κατάσταση ή η συγκεκριμένη πράξη εμπίπτει εντό ε, του ε, πεδίου του κοινοτικού δικαίου και επομένω και του χάρτη. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το ρόλο και του Οργανισμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και άλλων ενεξαρτήτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών διότι μπορούν να παρέχουν ενδείξει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι οποίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη της στα πλαίσια της παρακολούθησης από τα κράτη-μέλη για να ε, φροντίσουμε να εφαρμόζεται το νοσιακό δίκαιο και και ο χάρτης φυσικά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να προστατεύουμε τα δικαιώματα και των ε, ε, ατόμων. Μπορεί να υπάρχουν και μεμονωμένες καταγγελίες, διότι μπορεί για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση λόγω δικών της ερευνών, αλλά να λάβει υπόψη της και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία παρέχονται από πολίτες και βεβαίως ε, και ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων ε, για ε, τις μεμονωμένες παραβιάσεις τις οποίες δεν μπορεί να, στις οποίες μάλλον δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις συστημικού προβλήματος όσον αφορά ε, την συμμόρφωση της, ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και όλα αυτά φυσικά είναι και υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μία πτυχή όμως που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αναφέρουμε είναι η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη για τη μεταφορά ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας που έχουν σχέση με το χάρτη ώστε να είναι συμβατά με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ας πούμε μια εκ των προτέρων παρέμβαση προκειμένου να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν γίνεται μεταφορά της οδηγία θα γίνεται με τρόπο που θα συμμορφούνται και με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτή είναι μια πρακτική την οποία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας όπου η νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ε, κυρίως όσον αφορά την εξασφάλιση της αναλογικότητας ε, και την ε, συμμόρφωση των νομοθετικών παρεμβάσεων με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται λοιπόν για ένα προκαταρκτικό στάδιο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη τη και καλεί και άλλου ενδιαφερομένους ε, να ε, προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη του για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη ώστε να δουν πώ μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία με τρόπο που να συμμορφούνται πλήρω με το χάρτη. Και αυτό φυσικά έχει και κάποιες προεκτάσεις σε κάποιες περιπτώσεις τις οποίες ε, δίνονται και τομεακές κατευθυντήριες γραμμές από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή του χάρτη για την εκταμείευση ευρωπαϊκών κονδυλίων και από εκεί και πέρα σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προωθεί ε, τέτοια θέματα στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες ή συμμετέχουν στη διαδικασία της εκταμίευσης των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων Λοιπόν, αλλά φυσικά και ένα ακόμα παράδειγμα είναι ε, αυτά τα οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Δύο λόγια και για το τμήμα της στρατηγικής που αφορά την ευαισθητοποίηση. Να σας πω απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή σε εκπαίδευση, σε δημιουργία ικανοτήτων, πρώτων και κυριότερων εντός των θεσμικών οργάνων, δηλαδή επιμόρφωση για τους Ευρωπαίους ε, υπαλλήλους ε, ε, για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μάλιστα το τμήμα μου, το τμήμα θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων ε, και πολιτική θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Just παρέχει σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και επίσης εκπαίδευση για τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες σε εθνικό επίπεδο για την αποκεντρωμένη εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχές επιβολής του νόμου όσον αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά κυρίως ε, δικαστικούς και νομικούς για ε, ποινές και τη δικαστική εφαρμογή ε, του χάρτη. Έγινε ήδη μνήμα στην ετήσια έκθεση, όπως επίσης και η πρωτοβουλία που προωθεί ο πρώτος αντιπρόεδρος Τίμερμονς και η Επίτροπος Γιούροβα κάθε χρόνο να υπάρχει μια ετήσια συζήτηση για επίκαιρα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής και μάλιστα παρέχει και την δυνατότητα να ε, υπάρχει και συνέχεια με συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα μετά από τις συζητήσεις και στήριξη στους ενδιαφερομένους ε, και οργανώσει κοινωνία των πολιτών για τα θέματα που συζητούνται και πράγματι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών είναι ένα τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή είτε μέσω άτυπης, είτε μέσω πιο επίσημου και διαρθρωμένου διαλόγου, αλλά και δημοσίων διαβουλεύσεων και βεβαίως και οικονομικής ε, στήριξης. Ανέφερα στην αρχή ότι θα έλεγα και δύο λόγια για τα επιτεύγματά μας και τις προκλήσεις μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να έχουμε κάποια συνέχεια ε, μετά από αυτό το ισχυρό πλαίσιο και τη μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει στην εφαρμογή του χάρτη εντός των θεσμικών οργάνων και να δώσουμε τη δυνατότητα σε υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες να τα εφαρμόζουν όλα αυτά με ορθό τρόπο ε, και φυσικά να έχουν και τα σωστά αντανακλαστικά ώστε να αντιδρούν γρήγορα. Όλα αυτά, όπως είπα, γίνονται μέσω ε, εκπαίδευσης ε, προς τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τομεακά θέματα και τομείς πολιτικής στους οποίους είναι αρμόδια κάθε γενική διεύθυνση αλλά επίσης να προσπαθούν να αναπτύξουν και λίγο και να ενισχύσουν και τις δυνατότητες να παρακολουθούν τις τάσεις και να εξετάζουν και την εφαρμογή της νομοθεσίας επιτόπου και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Θα είδατε για παράδειγμα ότι σε πολλές από τις πρόσφατες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν συμπεριληφθεί και κάποιες γενικές διατάξεις στο τέλος που αφορούν την αξιολόγηση των μέσων που συχνά για παράδειγμα, αναφέρθηκα στην οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εφαρμογή της νομοθεσίας στα θεμελιώδη δικαιώματα. Να μην σταματάμε λοιπόν στην άσκηση της εξουσίας μας να υποβάλουμε προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα να εξετάσουμε και πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία επιτόπου και να γίνεται και μια αξιολόγηση εκ των υστέρων. Θα σταματήσω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πάρω εγώ το λόγο ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές, κυρίως τον καθηγητή Ντεσούτερ για την πολύ πολύτιμη μελέτη που μας παρουσίασε. Τα όσα κάνω οφείλουν πάρα πολλά σε αυτή τη μελέτη και το πρώτο αποτέλεσμα είναι αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε γιατί είναι στη διάθεσή σας, δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή ε, το δίνει η Επιτροπή εδώ σε κείμενο. Η σημερινή συντάντηση αποτελεί μια πρώτη ευκαιρία για να δώσουμε και το ενακτήριο λάκτισμα για την έρευνα ε, που πρέπει να προηγηθεί της κατάρτισης της έκθεσης. Και θα ήθελα λοιπόν επί τη ευκαιρία να θέσω κάποιες ερωτήσεις, κυρίως ε, όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα σημεία για τη σχέση της Ένωσης με το χάρτη. Σημεία τα οποία αφορούν κυρίως δύο θέματα. Τη δυνατότητα της επέκτασης της ερμηνείας του άρθρου 51 και το ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν άλλες πηγές δικαίου όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε, ο Κοινωνικός Χάρτης, ε, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ε, η Διεθνή Συνεργασία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά και τα Εθνικά Συντάγματα, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ράβο στην παρέμβασή της. Το παράδειγμα ε, το οποίο ε, προβάλλει περισσότερο την αμφισημία του άρθρου 51 είναι η οικονομική διακυβέρνηση που είναι προφανής ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τρόπον την είναι και ε, αδιαπέραστη ε, όσον αφορά τα όσα προβλέπει ο χάρτης. Όλα αυτά ξεκινούν από ένα όργανο το οποίο δεν είναι κοινοτικό, αλλά είναι διεθνές. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Σταθερότητας, όπως πολύ σωστά εξήγησε ο καθηγητής Δεσούτερ. Κάτι το οποίο δυσχεραίνει και την συμμόρφωση με το χάρτη. Υπάρχουν όμως οι φύνοντες σε πρώτο επίπεδο ε, και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν ουσιαστικά για τον Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό Σταθερότητας είναι δύο όργανα τα οποία είναι ε, πολύ σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και επομένω, και τα δύο, επειδή είναι θεσμικά όργανα της Ένωση, πρέπει να δρούν βάση του κοινοτικού κεκτημένου και επομένω πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τι επιταγές του χάρτη ε, που αφορούν και τις πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις πολιτικές εφαρμογής που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, μηχανισμέ, πολιτικές εφαρμογής οι οποίες είναι εγγεγραμμένοι ε, ε, στο ε, μνημόνιο συνεννόησης. Πρέπει δηλαδή τα μνημόνια να έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και όσον αφορά τα όσα προβλέπονται από το χάρτη, έχουμε αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κυρίω όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Ο καθηγητή Ντεσούτερ πολύ σωστά αναφέρθηκε στην ε, απόφαση Λίδρα Advertising ε, του 2007, που αφορά ε, το ε, μνημόνιο το οποίο υπεγράφει με την Κυπριακή Δημοκρατία και εκεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε σαφέστατα ε, ότι ισχύουν οι διατάξεις του χάρτη όσον αφορά τα θεσμικά όργανα και στις περιπτώσεις στις οποίες τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δρούν εκτός ενωσιακού πλαισίου. Αυτό το οποίο θα ήθελα να γνωρίζω είναι ποια είναι η οδός ώστε να γίνει ε, θεσμική μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 51. Το παράδειγμα το οποίο σας έδωσα για την απόφαση Λίδρα ε, του 2016 είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ε, στις αποφάσεις του δικαστηρίου και επομένως το δικαστήριο είναι πάρα πολύ περιοριστικό και εξετάζει την ερμηνεία του άρθρου 51 με πολύ περιοριστικό πέτρο, ε, τρόπο ή ε, το αντίθετο. Η καθηγήτρια Σπαβέντα, για παράδειγμα, λέει ότι το δικαστήριο είναι πάρα πολύ περιοριστικό όσον αφορά το άρθρο 51. Μια επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω, η δεύτερη ερώτηση, αφορά τι γίνεται με το χάρτη όταν ε, ε, οι ε, δράσεις έρχονται από το Eurogroup. Την ερώτηση την έφησε ήδη η πρόεδρος Χούμπνερ. Αλλά το παράδειγμα του Eurogroup είναι πολύ σημαντικό για όλες τις πολιτικές οι οποίες ε, θα αποφασιστούν στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Και εγώ φοβάμαι ότι θα γεννηθούν μια σειρά από οργανισμοί ενισχυμένης συνεργασίας που θα είναι στην πραγματικότητα διεθνείς συμφωνίες και επομένω δεν θα υπόκεινται στο χάρτη και κυρίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Ο καθηγητής Ντεσούτερ εξηγεί στο κείμενό του ότι οι διατάξεις του άρθρου 263 της συνθήκης όσον αφορά την ακύρωση δεν ισχύουν για το Eurogroup. Και επειδή το Eurogroup είναι ανεπίσημο όργανο, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις ε, ε μάλλον μπορεί να λάβει αποφάσεις που δεν έχουν ε, νομική υπόσταση. Και ε, εγώ θα ήθελα να ξέρω μήπως το Eurogroup θα μπορούσε ίσως να υπόκειται στο άρθρο 263 ως όργανο το οποίο περιλαμβάνεται στις συνθήκες. Άρα θα έπρεπε να υποβάλλεται στον έλεγχο της συμβατότητας με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως και τα υπόλοιπα όργανα. Επόμενη ερώτηση για τις άλλες πηγές δικαίου. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε στις αξιολογήσεις επιπτώσεων των διαφόρων οργάνων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε τη βαρύτητα των δικαιωμάτων που έρχονται να προσθεθούν ε, στα όσα είναι δεσμευτικά ε, συνταγματικά λόγω του χάρτη ο κοινωνικός χάρτης και άλλες πηγές δικαίου που αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να ξέρω. Δεν ξέρω μήπως ζητάω και πολλά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο χάρτη μεταξύ ε, πολιτικών δικαιωμάτων και ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Αναφέρεται και στη μελέτη του καθηγητή Ντεσούτερ, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι οι κοινωνικές αρχές δεν είναι τόσο δεσμευτικές μου φαίνεται ε, όσο τα πολιτικά δικαιώματα και είναι πολύ πιο δύσκολο ε, να, τα να τις προβάλλουμε. Επίσης, πώς μπορούμε να αποφύγουμε ο σεβασμός ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του χάρτη να μην γίνει μια απλή προστίκη η οποία θα γίνεται από εκεί και πέρα συστηματικά, απλώς ε, ρητορικά, συστηματικά σε όλες τις πολιτικές που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Να τα προσθέτουμε. Η μετανάστευση, για παράδειγμα, Προφανώς ε, υπάρχει, ε, έχει προφανή παραβίαση των θεμελιώδων δικαιωμάτων και πάντα στον προγραμματισμό να γράφεται πάντα αυτό θα γίνει πάντα με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο στην ουσία δεν θα σημαίνει τίποτα εάν αυτός ο σεβασμός δεν γίνει κάτι αυτόνομο και όχι απλώς ε, ένα κόμμα, μια υποδιαστολή που βάζουμε στο τέλος για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ικανοποιούνται με τόσο εύκολο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, συγγνώμη, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπροκ που δεν είναι εδώ, είναι σκιώδης συζητητές. Η κυρία Κάφμαν, καλημέρα. Έχετε το λόγο, είστε και εσείς σκιώδης συζητήτρια. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Μπάρμπαρα. Η σημερινή μέρα είναι μέρα όπου γίνονται πολλά ταυτόχρονα και γι' αυτό δυστυχώς ε, έχασα την αρχή της ε, συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συντάκτες της μελέτης. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική και σημαντική μελέτη που Ρίτα; επισημαίνει ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύει για όλους τους πολίτες ε, της Ένωσης ε, και είναι μεγάλη σημασίας όλοι οι αρμόδιοι, οι νομοθέτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα και φυσικά τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τον χάρτη σε ό,τι κάνουν. Τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχάς, διάβασα με ενδιαφέρον όσα αναφέρονται στη μελέτη για την οικονομική διακυβέρνηση. Βρίσκω σημαντικά και τα συμπεράσματα της μελέτης. Δηλαδή, όλα τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για να βγούμε από την οικονομική κρίση και κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο Ε, όσον αφορά λοιπόν αυτά τα εργαλεία βλέπουμε ότι δεν ε, έχει γίνει σεβαστός ο χάρτης στο σύνολό του. Πρόκειται για μια εκτίμηση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω διότι δεν επιτρέπεται σε κάποιους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, για παράδειγμα την ε, μακροοικονομική μεταρρύθμιση, δεν επιτρέπεται λοιπόν σε κάποιους τομείς ε, να μην εφαρμόζεται ο χάρτης. Άλλωστε είναι και προς όφελος των πολιτών, διότι για δικά τους δικαιώματα πρόκειται. Δεύτερη παρατήρηση, οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτοί παίζουν ρόλο σε σχέση με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι Οι εργασίες τους αφορούν 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με το συμπέρασμα που αναφέρεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στους οργανισμούς. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. και ίσως θα πρέπει να εκπονηθούν ε, περαιτέρω οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Άλλη παρατήρηση που δυστυχώς ε, δεν ε, λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στη συζήτησή μας είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τον χάρτη όταν εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο. αλλά το ερώτημα είναι σε τι βαθμό αποτελεί ο χάρτης κατευθυντήριο νήμα σε εθνικό επίπεδο. Και ιδιαίτερα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και οι εθνικές διοικήσεις, οι κυβερνήσεις φέρουν μεγάλη ευθύνη. Θα είναι λοιπόν χρήσιμο εάν προσέξουμε περισσότερο την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, στο εθνικό δίκαιο. Κυρία Ισηγήτρια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα πάνω στο θέμα αυτό καθώς και για το έγγραφο εργασίας που έχει δημοσιευτεί. Ελπίζω από κοινού να μπορέσουμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και προσβλέπω στη συνέχιση της καλής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σιλβί. Θα σας παρακαλούσα να είσαστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας, όχι παραπάνω από δύο λεπτά, διότι αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε τις απαντήσεις των ομιλητών μας. και του καθηγητή Ντεσχιούτερ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Ντόσκι. Όχι. Στην κυρία Μάιτε δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μας φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε και στις παρουσιάσεις αλλά και στα όσα μας παρουσίασε η Μπάρβαρα μέσω του δικού της έγγραφου και πρέπει να παραδεχτώ πως εδώ θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα ενισχύσουμε εμείς την ε, συμμόρφωση με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και αυτό θα αποτελεί ένα προηγούμενο βήμα πριν δημιουργήσουμε ε, την Κάρτα Ευρωπαίου ε, Πολίτη. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι ζωτική σημασία για εμάς και Παρόλο που ξέρω πως αυτό ακόμα δεν είναι πρακτικά εφικτό, νομίζω ότι αποτελεί ένα όνειρο κάποιων συναδέλφων και προς αυτή την κατεύθυνση θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν Μπάρμπαρα για τα όσα ε, μας βοήθησες να ακούσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ Μάιτε. Ο Γιώζεπ είναι ο επόμενος ομιλητής. για να σας πω ποια είναι η άποψη της Επιτροπής Αναφορών και μην ανησυχείτε να σας πω πως είναι οκτώ σημεία τα οποία μας ε, ανησυχούν, τα οποία είναι πολύ σύντομα. Λοιπόν, Πρώτον, ένα ε, σημαντικό αριθμό αναφορών που φτάνουν στην Επιτροπή μα οδηγούν σε να πιστεύουμε πω υπάρχει έλλειψη στην προσέγγιση ε, τη πολιτική ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτη-μέλη στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεύτερον, το πλαίσιο για τα θεμελιωδή δικαιώματα έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία, αλλά παραμένουν ακόμα μεγάλε διαφορέ ε, με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε στην πράξη. Τρία. Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε ε, την ισχύ υψηλών επιπέδων ε, σεβασμού των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων σε προηγούμενο στάδιο όλων των πολιτικών και νομοθετικών μας προσπαθειών. Τέσσερα, μας λυπά ιδιαίτερα η έλλειψη οποιασδήποτε διαβούλευση για τα θεμελιώδη δικαιώματα τη στιγμή που γίνεται η νομοπροπαρασκευαστική προετοιμασία των νομοθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει αυτό το θέμα να σε αυτό το θέμα να βελτιωθούμε. Πέντε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναθεωρήσουμε ε, το, τη συνέχεια που θα δώσουμε στο ECI. Δεύτερον, ε, έκτον, με συγχωρείτε, μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι κάποια κράτη-μέλη αδιαφορούν για τις υποχρεώσεις τους να ε, εξασφαλίσουν την εφαρμογή των θεμελιωδών και των μας λεπάει ιδιαίτερα η έλλειψη κοινοποίηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων προ του πολίτε και ο χώρο που δίνουμε στην κοινωνία των πολιτών, στον πολιτικό διάλογο που γίνεται δημόσια ε, και ο οποίο δεν είναι ε, αρκετό και τον οποίο δεν θα πρέπει να πιέζουμε ούτε με οικονομικού τρόπου ούτε με πολιτικού τρόπου. Και το τελευταίο και όγδο υπενθυμίζουμε τον τεράστιο ρυθμό αναφορών για το άρθρο 51 ε, το οποίο λαμβάνει η Επιτροπή μας και να σας πω πως τα άρθρα αυτά χρειάζονται ε, μια πιο ευρία ε, ερμηνεία, θέμα το οποίο πιέζει. Εσείς αναφερθήκατε σε μια εξαίρεση προηγουμένως, αλλά αγαπητοί Πρόεδρε, οι εξαιρέσεις δεν επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εσείς είπατε ότι η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αυτός είναι ο συνήθις τρόπος να τα λέμε. Δεν επιβεβαιώνουν τους κανόνες, αλλά απλώς αποδεικνύουν ότι οι κανόνες δεν είναι οι κατάλληλοι, διότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Ευχαριστώ. Μα, αυτή είναι η σημασία της εξαίρεσης που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Η η καλή εξαίρεση επιβεβαιώνει την ύπαρξη κακού κανόνα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Το, αυτή είναι η σημασία. Και τώρα... Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Α, ο κύριος Γιόγκ μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι εδώ μόνο ως εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Έχω δύο ερωτήσεις μία για τον καθηγητή κύριο Ντεσούτερ και να σας πω ότι πραγματικά με ε, κίνησε την περιέργεια το όσο είπε για την ε, διάσταση των εξωτερικών σχέσεων και πραγματικά όταν συνάψει κανείς μια εμπορική συμφωνία ή κάποια άλλη συμφωνία για να είναι πιο δραστήρες οι εμπορικές μας επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν θέματα που προκύπτουν για παράδειγμα η ΣΕΛ στην Ιγυρία για παράδειγμα επίσης εργασία των παιδιών οπότε Πρέπει να το δούμε αυτό και θα ήθελα να μου πείτε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε για τα θύματα που υπάρχουν σε τρίτες χώρες και που ζητούν ε, την εφαρμογή ένδικων μέτρων προστασίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ε, κενό και αυτά τα θύματα δεν έχουν δικαίωμα τέτοιου είδους προστασίας. Επίσης και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάβασα και άκουσα με ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα εσείς προσπαθείτε να κάνετε. Αλλά υπάρχει και μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που θα ζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στην Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού και το ελεγκτικό συνέδριο είδε πως υπάρχουν κάποιες πτυχές, κοινωνικές πτυχές στο πρόγραμμα στήριξης Ελλάδας που δεν έλαβαν καθόλου υπόψη το θέμα αυτό. Και μόνο που τώρα που γίνονται οι επιπτωσιολογικές μελέτες εξετάζεται αυτή η διάσταση και βέβαια είναι καθυστερημένο γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές μικρομεσαίες έχουν καταστραφεί, έχουν χρεοκοπήσει, έχει αυξηθεί η φτώχεια στην Ελλάδα και επίσης η Ελλάδα Ε, καταδικάστηκε και από το Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι η υποπτεύουσα αρχή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας. Οπότε εσείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνετε υπόψη αυτή τη χάρτα τη στιγμή που συνάβετε σχέσεις ή επιβάλλετε κάτι σε ένα κράτος μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ, Ντένις. Ε, ο κύριος Σεφλίν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. να ε, σας ευχαριστήσω για τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Ε, να σας διαβάσω κάτι. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απρόσβλητη, πρέπει να προστατεύεται. Αυτό είναι το άρθρο 1 του χάρτη ε, θεμελιωτών δικαιωμάτων. Αναφέρεται λοιπόν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αναφέρονται και οι οικουμενικές ε, αξίες ε, στο προήμιο και το άρθρο 2 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Κανείς δεν την ανέφερε. Γιατί? Τι ρόλο παίζει? Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να θεωρείται βασική αρχή όλων των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Καθηγητή της Πώς το βλέπετε αυτό και στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς έχει εφαρμόσει την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε τι βαθμό αποτελεί το μέτρο για όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα τους προσκεκλημένους μας ε, να παρέμβουνε και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολυάριθμες και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε πέντε από αυτές πολύ σύντομα, το υπόσχομαι. Κυρία Σπινέλη, Ρωτήσατε σχετικά με πηγές άλλες από τον ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Νομίζω ότι είναι σημαντικές πηγές που η συνθήκη στο άρθρο 6.3 απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη πέρα από τον χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων. Ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είχε σκοπό να παγώσει το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η μόνη πιο σημαντική πηγή που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη είναι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικό Χάρτης. Γιατί? Διότι, καταρχάς, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει επιλέξει κάποια στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και δεύτερον, βλέπουμε αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το πώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο, χάρτης, ε, ο κοινωνικός χάρτης ε, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ο, και το σώμα των εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν την εφαρμογή του χάρτη θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνεται υπόψη στην νομοθεσία και έχουμε την ε, υπόθεση Confederation Générale du Travail κατά της Γαλλίας του Ιουνίου του 2010. Όπως γνωρίζουμε, μετά την απόφαση Λαβάλ του δικαστηρίου στις 18 ε, Δεκεμβρίου του 2017, ο Σουηδός νομοθέτης τροποποίησε το δίκαιο της Σουηδίας λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή. Και αυτό οδήγησε στο να θεωρηθεί ότι η Γαλλία είχε παραβιάσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη σε μια υπόθεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Σουηδίας. Και έχουμε διάφορες αποφάσεις ε, φυσικά που αφορούν την Ελλάδα που θεωρούν ότι η Ελλάδα παραβιάζει τον ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη παρότι η Ελλάδα απλά εφήρμοζε τα μνημόνια του 2010 και του 2012. Το πιο σημαντικό μήνυμα εδώ λοιπόν είναι ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι πλήρης όσον αφορά τις παραπομπές ε, και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το άρθρο 6.3 και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Κυρία Σπινέλη, αναφερθήκατε στο Eurogroup. Όταν το Eurogroup παίρνει θέση, πρόκειται για πολιτική θέση, η οποία κατόπιν εφαρμόζεται με μέτρα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Και έχουμε την ε, περίφημη υπόθεση της Ledra Advertising, όπου το Eurogroup είχε επικροτήσει μία απόφαση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Κύπρο. Και κατόπιν αυτής της ευλογίας ε, ε, του Eurogroup ε, η Κύπρος εφήρμοσε μέτρα τα οποία κατόπιν διαπιστώθηκε ότι αντίκειται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Eurogroup λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ότι ό,τι απόφαση και να πάρει πρέπει να συμμορφώνεται με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι αλλιώ εκ των υστέρων θα υπάρξουν συνέπειε. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό συμπέρασμα ε, τη υπόθεση ε, Letter Advertising του Δεκεμβρίου 2016. Άλλη ερώτηση για τα κράτη-μέλη που έθεσε ε, Ευρωβουλευτής της Επιτροπής σας. Τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν καλύτερη καθοδήγηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για οδηγίες, στην περίπτωση των οποίων τα κράτη-μέλη έχουν σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή τους. Οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών ανησυχούν ότι οι οδηγίες δεν είναι αρκετά ακρίβεις σχετικά με το τι μέτρα δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να λάβουν τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή τους. Και σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να βοηθά τα κράτη-μέλη. Και το ίδιο ισχύει για τον Οργανισμό Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Και χάρηκα πολύ που η κυρία Χάβο αναφέρθηκε στην εκ των υστέρων αξιολόγηση των ε, νομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα τι κάνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή. Επίσης πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν περισσότερο για να ενισχύσουν τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δικαιοδοσίε των κρατών μελών αποτελούν ε, μέρος ενός ενιαίου δικαστικού συστήματος και είχαμε την υπόθεση του 1986 Λεβέρ κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, πρέπει να προστατεύεται το κράτος δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά ε, στην ε, νομική προστασία. Και αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη δεν κάνουν ε, όσα θα έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο 19 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Τερικάπρας από την Επιτροπή Αναφορών είχε κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία από αυτές. Ε, δυστυχώς έχει εγκαταλείψει την αίθουσα, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πολλές από τις αναφορές που καταλήγουν στην Επιτροπή Αναφορών αποτελούν ε, πηγή πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πιθανές διαδικασίες επιπαραβάση κατά κρατών μελών που παραβιάζουν ε, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, σχεδόν απεριόριστο, όσον αφορά την προσφυγή κατά κρατών μελών. Ε, εγώ θα πρότεινα, αφού η, Επιτροπή Αναφορών εξετάσει μια αναφορά, ακούσει τις ανησυχίες των πολιτών, να επιβάλλει στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιπλέον υποχρέωση να δικαιολογήσει σε περίπτωση που δεν προσφύγει κατά κάποιου κράτους μέλους στην περίπτωση αυτή τα πολιτικά παζάρια εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όταν ε, επιλέγει κατά ποιον κρατών θα ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση είναι θέμα που προκαλεί ανησυχίες. Και όσον αφορά τον κύριο Δεγιόν από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, σχετικά με τρίτες χώρες, ε, πράγματι είναι σημαντική η ανησυχία του. Έχουμε κανονισμό, τον κανονισμό Βρυξέλλες 1, 44 κάθετος 2001 που επιτρέπει σε ε, θύματα ε, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ε, ευρωπαϊκές εταιρείες σε τρίτες χώρες μπορούν να προσφύγουν στο κράτος μέλος της επιχείρησης. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται πιο συστηματικά και θα πρέπει να διευκολύνουν τα κράτη-μέλη την πρόσβαση για τα θύματα σύμφωνα με αυτά που ε, έχει πει στην παρατήρηση παριθμών 24 η ε, ε, Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί αναφέρεται ότι υπάρχει υποχρέωση διευκόλυνση από πλευρά των συμβαλωμένων μερών. Και όλα τα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει αυτό το σύμφωνο. Δυστυχώ όμω στι παρούσε συζητήσει για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει πολύ αμυντική θέση εντός του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με νέα συνθήκη πάνω στο θέμα αυτό, παρότι η Επιτροπή θα ήθελε να δημιουργήσει συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, ώστε όλες οι περιφέρειες του κόσμου να παρακολουθούν προσεκτικά τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους, όπου και αν ε, αυτές επιχειρούν. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στις κάτω ε, Τον Μάρτιο του 2016 είχαμε την αυτή νομοθεσία στη Γαλλία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια, που αποτελεί ένα χρήσιμο πρόσθετο εργαλείο. Ε, επιχειρήσεις λοιπόν που δεν ε, γνωρίζουν ποιες ε, είναι οι υποχρεώσεις τους ε, και λόγω των ε, στρεβλώσεων στην αγορά πιστεύω ότι στον τομέα αυτόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας παρουσιάσω λοιπόν και την άποψη της Προεδρίας. Τώρα σχετικά με την οικονομική διάσταση και το θέμα που θίξατε. Όπως και με όλες οι υπόλοιπες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή ε, της χάρτας, οπότε ναι, πρέπει να εφαρμόζεται στο 100% και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για την ε, υπηρεσία. Να σας πω πως ε, ναι, καλή ιδέα το να αυξήσουμε την ε, ορατότητα αυτής της υπηρεσίας, να έχουμε μια μεγαλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τα σχετικά σας σχόλια σαφέστατα, ε, έχετε δίκιο, θα πρέπει να θεωρούμε ότι παίζει ένα κρίσιμο ρόλο. Τώρα για τα κράτη-μέλη, βεβαίως και αυτά υποχρεούνται στο να εφαρμόζουν την ε, χάρτα όταν εφαρμόζουν ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και βεβαίως Ξέρουμε, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πως τα δικαστήρια όλο και περισσότερο αναφέρονται σε αυτή τη χάρτα στις αποφάσεις τους. Τώρα, το τι συμβαίνει όταν κάποια κράτη-μέλη ε, αγνοούν ε, τα δικαιώματα αυτά. Νομίζω ότι αποτελεί μια κοινή ευθύνη να υπενθυμίζουμε στους αυτούς μας ποια είναι τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και βεβαίως ο θεματοφύλακας των συνθήκων αντίστοιχα μπορεί να το πράξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με την Κομισιόν και με άλλους ομιλητές πως υπάρχουν και άλλε πηγές νομοθεσία σχετικέ με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει και αυτές να λαμβάνονται υπόψη και εδώ να φέρουμε πιο συγκεκριμένα στην ύπατη αρμοσία, όπως επίσης και στο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη ε, να αποτελέσει και αυτή τη μήμα αυτής της σύμβασης. Έχουμε τα άρθρα 53 εδώ της χάρτας για παράδειγμα που ε, περιγράφει πολύ σωστά πως οι διεθνείς συμβάσεις δεν περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θέλετε κι εσείς να πάρετε το λόγο? Ναι. Μικρόφωνο παρακαλώ. Θα απαντήσω ε, στα, γρήγορα σε τέσσερα σημεία. Να σας πω πως ακούστηκε μία ερώτηση από τον κύριο Ντεγιόγκ για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και το πώς οι κοινωνικές διαστάσεις δεν ελήφθησαν υπόψη επαρκώς ε, στο μνημόνιο ε, και στο σχετικό πρόγραμμα για την Ελλάδα να σας πω εκ μέρους εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για οποιοδήποτε μελλοντικό πρόγραμμα αντίστοιχο και βεβαίως αυτοί οι προβληματισμοί θα ληφθούν υπόψη ε, στις ε, σκέψεις που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κοινωνικό πυλώνα. Δεν είμαι σε θέση να δώσω αυτή τη στιγμή παραπάνω λεπτομέρειες. Για την ε, επιβολή και για τις ε, ε, αναφερθήσεις παραβιάσεις από πλευρά κρατών μελών. Ε, θα επαναλάβω πως εμείς συμφωνούμε σίγουρα όλοι με το γεγονός πως ε, η εξέταση της εφαρμογής στην πράξη θα πρέπει να γίνει με, παράλληλα με μια εξπόστα αξιολόγηση των βασικών εργαλείων και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη ανέφερα και νομίζω ότι και ο καθηγητής κ. Ντεσούτερ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Τώρα, για τις αναφορές, ναι, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις αναφορές, τις αναλύουμε εντελεχέστατα, αναμφίβολα, και όταν έχουμε τέτοιου είδους ενδείξεις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού ε, νόμου ε, το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Συχνά συμβαίνει οι αναφορές να θέτουν θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της χάρτας. Οπότε εδώ ίσως χρειάζεται και συνεργασία έτσι ώστε να φιλτράρονται οι αναφορές. Ίσως και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και για τις παρεμβάσεις εκ των προτέρων, εξάντε, από τα κράτη-μέλη τη στιγμή τη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και το κατά πόσο συμμορφώνονται με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θα μιλήσω για τα σεμινάρια αυτά μεταγραφή ε, και μάλιστα να σα πω πω η Υπηρεσία Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων έχει εμπλακεί πολύ δραστήρια με πολύ πολύτιμη συμβολή και εδώ θα πω πως ε, συμμετέχουν και στην ε, πολύ συχνά στην, σχεδόν πάντοτε θα έλεγα στην διατύπωση των νομοθετικών προτάσεων ε, όταν βέβαια ε, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη και στις εσωτερικές ομάδες εργασίας όταν προκύπτει κάποιο θέμα πάντοτε τώρα η κοινωνία των πολιτών Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως βεβαίως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ένας πολύ πολύτιμος σύμμαχος στην προστασία των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο ρόλος τους. Έχουμε ε, δεσμευθεί πως θα τις στηρίξουμε τις οργανώσεις αυτές με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ε, αυτό το χώρο που όλο περιορίζεται, το shrinking space με μία έρευνα που έχουμε ξεκινήσει για το σχετικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παρουσιαστεί και η σχετική έκθεση το Δεκέμβριο και τα αποτελέσματα θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε μέσω μιας πιο εις βάθος μελέτης έτσι ώστε οι κοινωνίες των πολιτών ε, να στηριχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κατάλληλο τρόπο. Τώρα για τις νομοθετικές εξελίξεις και την διαχείριση που γίνεται σε εθνικό επίπεδο που μπορεί να περικόπτει τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανωτικών οργανώσεων με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ε, ε, παρακολουθούμε. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες με παραβάση κατά της Ουγγαρίας για παράδειγμα και είμαστε σε διάλογο με την χώρα αυτή για να διαπιστώσουμε αν αυτή η παραβίαση ε, της χάρτας και του ευρωπαϊκού δικαίου μπορεί να, να ξεπεραστεί. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές και ελπίζω να μείνουμε σε επαφή. And now... Ε, και τώρα... Περνάμε στο επόμενο σημείο. Η εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης ε, για τα Εθνικά Κοινοβούλια κύριος ε, Πάλο Ραγγέλ, είναι ο εισηγητής. Ανέλαβε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2016 καθήκοντα για αυτή την ε, έκθεση εφαρμογής και αυτούς τους μήνες ε, έκανε διάφορες συλλεκτικές δραστηριότητες, είχαμε εργαστήρια, ε, αποστολές διερευνητικές, αξιολογήσεις επιπτώσεων, ε, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σήμερα θα περάσουμε απευθείας στην εξέταση του σχεδίου έκθεσης βάσει και των ε, διατάξεων όσον αφορά τις, εκτελεστικές, ε, τις εκθέσεις εφαρμογής θα πρέπει να εγκριθούν σε επίπεδο επιτροπής εντός ενός έτους από την έγκριση εκτός ε, και αν υπάρχει ε, ε, συγκεκριμένος λόγος, ο οποίος εγκρίνεται και από τους συντονιστές για παράταση. Για τη συγκεκριμένη έκθεση δόθηκε παράταση από τις 7 Ιουλίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2018, συγγνώμη, ζητήθηκε η παράταση και μετά από αυτή τη συζήτηση στην ΑΦΚΟ που έγινε στις 10 Οκτωβρίου ε, του εγγράφου εργασίας, ο εισηγητής, ο Παύλο Ρανζέλ, θα παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο εκθεσής του. Παρακαλώ, κύριε Ρανζέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια οργανωτικά. Νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την έκθεση στην ΑΦΚΟ τον Ιανουάριο, αλλά βεβαίως αυτό θα εξαρτηθεί και από και τις διάφορες θέσεις που θα παρουσιαστούν κυρίως όσον αφορά τις τροπολογίες. Βεβαίως αυτό εξαρτάται και από τη μετάφραση και την τεχνική αναθεώρηση η οποία υπολογίζω ότι θα γίνει αρκετά γρήγορα αλλά οψόμεθα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης και να εξετάσουμε και κάποιες τροπολογίες Κάποια πράγματα τα είδαμε και στο έγγραφο εργασία ήδη, αλλά τώρα σε επίπεδο τουλάχιστον επιτροπής ε, ε, και επίτροπο διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών πρέπει να τα παρουσιάσουμε διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουν άμεση σχέση και υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ε, συνδιοργανώνονται με τα Εθνικά Κοινοβούλια επομένως υπάρχει εμπειρία και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό επιπλέον και σε άλλες πλατφόρμες οι οποίες είναι λίγο πιο ανεπίσημες αλλά εδώ στις Βρυξέλλες ε, ε, έχουν εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων θα παρουσιάσουμε δηλαδή και εκεί το σχέδιο κειμένου πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθεί το έγγραφο και με αυτές τις οργανώσεις σε διάφορα επίπεδα ώστε να μην τα δούμε μόνο στην ατμόσφαιρα στο στο περιβάλλον εδώ της Επιτροπής μας. Πρακτικά τώρα οι προτάσεις που ήδη συζητήθηκαν όταν συζητήσαμε το έγγραφο εργασίας αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο έκθεσης παρόλο που νομίζω ότι προσπαθεί να προσδώσει ένα θεσμικό πλαίσιο, συνταγματικό μάλλον πλαίσιο, με μια πιο καινοτόμα προσέγγιση για τη συμβολή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ξεκινούμε λέγοντας το προφανές ε, και στην παράνθεσή μας έχουμε τις εκθέσεις Ναπολιτάνο, Καζίνη, Μπρόκ κλπ. Και αυτό είναι ότι η βασική λειτουργία των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι να ελέγχει τη δραστηριότητα του ε, κυβέρνησης. Γιατί ε, στην κυβέρνηση ε, έχουμε εκπροσώπηση στο Συμβούλιο και φυσικά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν μέσα εργαλεία άσκησης ελέγχου στις εκτελεστικές εξουσίες. Αρχίζουμε λοιπόν ε, τονίζοντας τη βασική λειτουργία των Εθνικών Κοινοβουλίων και εδώ προσπαθούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Πρώτον, σε επίπεδο ΚΟΖΑΚ, ακόμα και σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, συζητήσεις για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σύγκριση βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να σας πω ότι στις επαφές μου και στις συναντήσεις μου με προσώπους των διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων πάντα ε, ζητούν ανταλλαγή εμπειριών στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν την εκτελεστική τους εξουσία, ε, οι, πώς λειτουργούν οι επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων σε εθνικό επίπεδο, εάν συναντιούνται με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ούτω καθεξής, αλλά επίσης ε, τι περιλαμβάνεται στον κανονισμό του σε εσωτερικό επίπεδο και τι σημαίνει αυτό, τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους, τι εργαλεία διαθέτουν προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν κάποια επιρροή ε, στα όσα κάνει η κυβέρνησή τους. Και φυσικά εδώ νομίζω ότι ε, έχουμε και μία από τις ουσιαστικές πτυχές, ε, παρά το γεγονός ότι είναι στην αρχή της έκθεσης, και εγώ θεωρώ ότι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υποστηρίζουμε λοιπόν ακράδαντα την ε, αναβάθμιση των δυνατοτήτων του IPEX. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο υποστήριξε ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και εγώ τολμώ ε, να αποκαλέσω αυτή τη πλατφόρμα ένα βήμα, μια αγορά ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανταλλαγή πληροφοριών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ου μόνον για να μπορούν να ασκήσουν το ρόλο τους στα εθνικά κοινοβούλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τον έλεγχο των εθνικών τους κυβερνήσεων, διότι μέσω του IPEX μπορούν να παρακολουθούν ποια θέματα συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα μπορούσε να ε, αποβεί πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ δε πηγαίνουμε και λίγο παραπέρα και αυτό ε, ήδη το συμπεριλάμβανα και στο έγγραφο εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό δηλώνοντας με πολύ επίσημο τρόπο ότι σεβόμαστε και το δικαίωμα κάθε κοινοβουλίου να αυτοδιοργανώνεται, να καθορίζει τον κανονισμό του και ε, αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι γερμανόφωνοι από τον όρο της ε, εξουσίας, ε, της δυνατότητας για αυτοοργάνωση που χρησιμοποιείται στα γερμανικά. Αρκετές φορές ακούσαμε ε, ε ισχυρισμούς εθνικών κοιτοβουλίων κατά του Ευρωπαϊκού Εξαμένου, γιατί λέει ότι αποδυναμ... λένε ότι αποδυναμώνεται η εξουσία του σε εθνικό επίπεδο μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξαμήνου. Αλλά αν εγκρίνουν κανονισμό ο οποίος ε, θα προλαμβάνει μεγάλο τμήμα της συζήτησης σε θέματα προπολογισμού, τότε διαθέτουν μέσα τα οποία μπορούν να του επιτρέπουν να ελέγχει το διάλογο μεταξύ κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ε, κυβέρνηση και Συμβουλίου σε όλα τα θέματα προπολογισμού και επομένω μπορούμε να έχουμε και ένα εθνικό ε, τρίμηνο, αν θέλετε, πριν από το ευρωπαϊκό εξάμεινο και μπορεί να παρακολουθούν εκεί όλες τις ανταλλαγές επόψεων και των θέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Κυβερνήσεων ώστε ορισμένες φορές αυτό που γίνεται το οποίο ε, φυσικά ε, σε κάποιο βαθμό αφορά μόνο τα εθνικά κοινοβούλια είναι ότι αν θέλουν να αλλάξουν τον ιστορικό τους κανονισμό έχοντας κατά νου ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο θα μπορούσαν να έχουν και τη δυνατότητα στη συνέχεια να έχουν μία επιστροφή των ε, ε, ε, εξουσιών προπολογισμού, κατάρτιση προπολογισμού που πίστευαν ότι έχουν στο παρελθόν και χάνουν τώρα. Πρέπει δηλαδή, κατά μία έννοια, να έχουμε μια παράλληλη διαδικασία μεταξύ των όσων συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των όσων συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να έχουν σημαντική βαρύτητα σε αυτά τα θέματα, σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ε, λειτουργία που είναι ο έλεγχος της κυβέρνησής τους, εάν προσαρμόσουν κατά το σωστό τρόπο τον εσωτερικό τους κανονισμό στις διαδικασίες που έχουμε στις Βρυξέλλες, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πρόταση απλή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το δηλώσουμε εδώ διότι υπάρχουν ε, αποτελεσματικές δυνατότητες ε, οι οποίες ε, μπορούν να επιτρέψουν την πλήρη σκή στα εθνικά κοινοβούλια εάν μπορούν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατόπιν υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Η συνθήκη της Λισαβόνας, προηγουμένως η συνθήκη του Άμστερνταμ, αλλά ιδίως η συνθήκη της Λισαβόνας, είναι η συνθήκη των κοινοβουλίων. έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ περισσότερες εξουσίες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν και αυτό είναι απόλυτα σαφές και υπάρχει και συγκεκριμένος ρόλος για τα Εθνικά Κοινοβούλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλέον λοιπόν δεν ε, έχουμε μόνο ρόλο εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τις κυβερνήσεις τους, αλλά και ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ ε, εγώ πάντα ε, θέτω στον εαυτό μου την εξής ερώτηση. Εάν τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί να έχουν λόγο τα εθνικά κοινοβούλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι μπορούν να κάνουν το οποίο είναι διαφορετικό. Προσπαθώ δηλαδή να ορίσω την συγκεκριμένη διαφορά, να χρησιμοποιήσω και το λατινικό όρο, differentia specifica, μεταξύ εθνικής κυβέρνησης και εθνικού κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι τα εθνικά κοινοβούλια προσδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εσωτερική ποικιλομορφία. Όταν η κυβέρνηση ψηφίζει στο Συμβούλιο, πρόκειται για μια αδιαίρετη ψήφο που εκπροσωπεί τη βούληση ενός κράτους αλλά είναι αδιαίρετη. Όταν όμω ένα κοινοβούλιο έρχεται εδώ σε μία συνεδρίαση, έρχεται μέσω εκπροσώπων και εκεί υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπηση διαφόρων απόψεων. Είναι παρούσα αυτή η διαφορετικότητα. Ορισμένε φορέ η μειοψηφία στη Σλοβακία μπορεί να είναι η πλειοψηφία στο Βέλγιο και η μειοψηφία στη Σουηδία να είναι η πλειοψηφία στη Μάλτα ή στη Γερμανία και μπορούν να έχουν αλληλεπιδράσεις. Ουσιαστικά δημιουργούν ε, μια πολιτική αρένα και μέσω της ειδική τους της ε, διαφορετικότητα συνεισφέρουν στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας διότι εκφράζουν το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην εθνική πολιτική σφαίρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο που είναι το επίπεδο του Συμβουλίου που ε, έχουμε τη βούληση του κράτους, αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, το επίπεδο των κοινοβουλίων, που εκφράζει και την πολυφωνία και τις διαφο διαφορετικές απόψεις και για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο εδώ προτείνουμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και μάλιστα κατά πολύ, διότι πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό, ε, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων σε όλες τις συνεδριάσεις να αντανακλούν και την πολυφωνία που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι καλό ότι οι πρόσφατες ε, απόψεις οι οποίες εκφράζουν με σαφή τρόπο την βούληση του Κοινοβουλίου ε, μπορεί να είναι και διστάμενες απόψεις. Δηλαδή να δίνεται χώρος στις μειοψηφίες να πούν γιατί διαφωνούν με κάτι συγκεκριμένο. Αυτό θα μπορούσε να είναι και συμβολή στην όλη διαδικασία ε, προσφοράς ε, στα εθνικά κοινοβούλια, να τους προσδώσουμε το ρόλο που τους αρμόζει. Αυτό βεβαίως γίνεται σεβόμενοι δύο πράγματα. Πρώτον, κατά πόσον υπάρχει ε, ε συγκεκριμένη άποψη της πλειοψηφίας, η ε, άποψη του Εθνικού Κοινοβουλίου είναι η άποψη της πλειοψηφίας. Αυτό είναι φυσικό. Δεύτερον, αυτό γίνεται μόνο εάν ο κανονισμός κάθε κοινοβουλίου το επιτρέπει, διότι πρέπει να σεβαστούμε και την ε, δυνατότητα αυτοοργάνωσης που έχει κάθε κοινοβούλιο. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες προτάσεις που ελπίζω ε, και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να δώσουν στα εθνικά κοινοβούλια και έναν αυτόνομο ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, βεβαίως, προτείνουμε και κάποιες απλουστεύσεις ε, όλων των συνοδριάσεων που έχουμε. Προτείνουμε, για παράδειγμα, διότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο με την ICM, με την Κόζα, έχουμε, Κόζα και έχουμε κοινέ συνεδριάσεις, έχουμε θέματα ασφάλειας και ελευθερίας, ε, την ε, ε, Αμυντική Ένωση κλπ. Και αυτά θα έλεγα πως είναι τα πλαίσια στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάποιο είδους πρότυπα. Δηλαδή, πιστεύω πως αυτή την διαδρομή θα έπρεπε να την εξερευνήσουμε, να δούμε εάν μπορούν μέσω αυτών των διαδικασιών να συμμετέχουν. Να πω παρεπιπτόντως πως σε μία ε, πρόταση που είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αλλά μπορεί να εφαρμοστεί είναι η Ευρωπαϊκή Οδός. Δηλαδή καλό θα ήταν να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που θα μπορούσαμε ταυτόχρονα σε όλα, τα 27 κοινοβούλια ταυτόχρονα να γίνεται μια συζήτηση, ένας διάλογος για τα ευρωπαϊκά θέματα. Θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα συζητιέται ή ε, κάποιες θεσμικές διευθετήσεις. Θα μπορούσε να είναι η αμυντική άμυνα. Και Και εδώ θα είχαμε τη συμμετοχή όχι μόνο των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά επίσης μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το λέω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μιλώ για τα ε, μέλη του Εθνικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το οικείο κράτος μέλος, αλλά αλλοδαπά ε, μέλη έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική ανταλλαγή, ένας πραγματικός διάλογος για τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Και ο τρόπος αυτός θα έδινε, αν θέλετε, ένα βαθμό πρακτικής εφαρμογής αυτής της ε, δημοκρατικής σύμβασης ε, στην οποία αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Μακρόν που ακόμα δεν είναι ακριβώς σαφές τι επιδιώκει αλλά κάτι, τέτοιο και τέλος και δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί έχω ήδη 15 λεπτά που μιλάω περίπου έχουμε επίση και τον έλεγχο επικουρικότητας είναι αυτό το οποίο προβλέπεται στο πρωτόκολλο ως βασικό εργαλείο. Και εδώ έχουμε ε, ε, ακούσει και διάφορα αιτήματα και αισθήματα εκνευρισμού από τα Εθνικά Κοινοβούλια πως δεν επαρκεί, πως οι 8 εβδομάδες θα έπρεπε να γίνουν 12 πως οι χρονικές προθεσμίες δεν είναι πολύ λειτουργικές, πως χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Αυτό όμως βρίσκεται ε, στην ε, συνθήκη και καταλαβαίνετε πως κάτι τέτοιο απαιτεί τροποποίηση αυτής. Αυτό το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε και νομίζω ότι είναι πράγματι εφικτό, είναι να ε, εντάξουμε μια τεχνική περίοδο μέσα σε αυτή την προθεσμία Οπότε να μην είναι στη διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια είναι η αρχή αυτής της διαδικασίας, αλλά να προβλέψουμε και κάποιες ημέρες τεχνικής ε, άδειας, έτσι ώστε όλα τα εθνικά κοινοβούλια να είναι σε θέση να λάβουν τα έγγραφα, να τα διαβάσουν, να τα κατανοήσουν στη γλώσσα τους και να έχουν πραγματική γνώση του τι συμβαίνει. Και αυτό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη δέχεται πως ο μήνας Αύγουστος δεν μετράει μέσα στην ε, περίοδο των 8 εβδομάδων γιατί συνήθως ε, βρίσκονται σε αργία οι... τα εθνικά κοινοβούλια οπότε Νομίζω πως εδώ μπορούμε να ανοίξουμε ένα περιθώριο και να δώσουμε και επιπλέον 5-6 μέρες για παράδειγμα για την κοινοποίηση, όπως έχουμε σε διάφορες εθνικές ε, διαδικασίες. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο ενδεχομένω θα δημιουργήσει περισσότερες ε, αντιμαχίες είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί πάντα το επιχείρημα της επικουρικότητας με μια πολύ περιοριστική και αυστηρή ερμηνεία. Ποιος διαβάζει το δημόσιο δίκαιο στην Ευρώπη. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Αγγλία. Ξέρετε πως η επικουρικότητα μπορεί να ερμηνευθεί αυστηρά. Και να πούμε πως ισχύει μόνο για τις πολιτικές αρχές που διακυβεύονται ή μπορεί κανείς πιο ε, διευρυμένα να θεωρήσει πως υπάρχει παραπομπή και αναλογικότητα. Εγώ λοιπόν λέω στην Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι λοιπόν λίγο πιο περιοριστική εγω λοιπον λεω στην ευρωπαικη επιτροπη ερμηνεύει την επικουρικότητα γιατί εγώ ως νομικός πρέπει να σας πω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να διακρίνει κανείς και να ορίσει τη γραμμή μεταξύ όσων ανήκουν στην επικουρικότητα και των όσων ανήκουν στην αναλογικότητα. Άρα λοιπόν, η κίτρινη κάρτα ουσιαστικά θανατώνεται με την υπερβολικά περιοριστική ερμηνεία της ε, επικουρικότητας γιατί δεν αφήνει χώρο καθόλου για την άσκηση αυτού του πολιτικού ελέγχου. Και εμείς λέμε ότι τα προβλήματα με την πορτοκαλί και την κίτρινη κάρτα δεν είναι μόνο προβλήματα χρονικών ε, προθεσμιών, αλλά και με την ερμηνεία του τι ανήκει πραγματικά στην αρχή της επικουρικότητας. Και επιτρέψτε μου και ένα ελάχιστο σχόλιο. Καμιά φορά ακούω τον κύριο Τίμερμαντς Μείωση νομοθεσία, ε, επιτροπές, απλούστευση τα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ερμηνεία τη επικουρικότητα, η οποία θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι πιο ευέλικτη, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα χρειαζόταν καν τέτοιου είδου προσπάθειε. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί, γιατί του αρέσει πάρα πολύ να μειώνουν την νομοθεσία, αλλά μετά όταν πάνε να ε, εφαρμόσουν την αρχή της επικουρικότητας, νομίζω κάνουν κάτι σχετικά διαφορετικό με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ράντζελ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εισαγωγή. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο τώρα στη διάθεσή μας. Θα είμαι λοιπόν πολύ αυστηρή όσον αφορά τον χρόνο ομιλίας των σκιωδών. Όχι παραπάνω από δύο λεπτά. Λείπαμε πάρα πολύ. Αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δίνω το λόγο στην κυρία Περβάνος Περέζ. Euh, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την αμέση εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια λοιπόν και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε αλλά χαίρομαι, χαίρομαι που κατάφερε ο συγητής να μας καταθέσει αυτή την πολύ λεπτομερή ε, εργασία από την στιγμή που ξεκίνησε η θητεία του εργάστηκε σκληρά και εξακολουθώ να πιστεύω πως το να περάσουμε από την Ολομέλεια τον Ιανουάριο είναι υπερβολικά αισιόδοξο σενάριο αλλά θα προσπαθήσουμε, θα δουλέψουμε σκληρά και νομίζω ότι θα είναι το σωστό timing γιατί τελικά το θέμα το οποίο έχετε βάλει εσείς στην έκθεσή σας εντάσσεται σε μια γενικότερη ευρύτερη συζήτηση που είναι ποια είναι η επίπτωση και η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία σημεία στα οποία αναφερθήκατε εσύ και θα σταθώ εγώ. Οι περιορισμοί για τα εθνικά κοινοβούλια. Ναι, έχουμε μια ιστορική δυσκολία την οποία γνωρίζουμε και η οποία θα μας οδηγήσει στο να, να δώσουμε περισσότερα κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχει ε, μια ευρωπαϊκή δυναμική η οποία ε, θα τους επιτρέψει να δουλεύουν πιο σκληρά. Αλλά τώρα το νέο ε, το νέο αυτό, οι νέες προθεσμίες ε, που προτείνεται θεωρώ πως δύσκολο ε, θα φέρουν θετικά αποτελέσματα είναι υπερβολικά και αυτές περιοριστικές. Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα είναι αυτό που είπαμε συνέλευση. Δεν το είπαμε ακριβώς συνέλευση, αλλά είναι αντίστοιχο με αυτό που ολομέλεια περιουσιάζετε εσείς. Σίγουρα θα έχει επίπτωση γιατί υπάρχουν τα θέματα της άμυνας, υπάρχει το θέμα της ΟΝΕ, ναι, υπάρχει ο τρίτος πυλώνας, οπότε θα μπορούσαμε ναι, να τα συνδυάζουμε με αυτά τα οποία συζητούν στα Εθνικά Κοινοβούλια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τις μοιρασμένε εισαγωγικά αρμοδιότητες και ίσως αυτό όμως αν προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε μας δημιουργήσει πρόβλημα στο πώς θα τα συνδέσουμε μεταξύ μας. Τώρα για την ε, συνέλευση τι είναι αυτές οι συνελεύσεις ε, πολιτών και πώς μπορούν αυτές να συνδυαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Εθνικό Κοινοβούλιο. Ε, πώς μπορούν λίγοι να γίνουν αυτές οι σκέψεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τρόπο που περιγράφεται. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ερωτήματα στα οποία θα κληθούμε να απαντήσουμε. Κύριε θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Θα είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις συστάσεις στην έκθεση του κυρίου Ρανζέλ. Και αυτές που αναφέρονται στη πιο αυστηρή ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας. θα πρέπει να έχουμε σχετικά ευέλικτο σύστημα ώστε να έχουμε εγκαίρως τη θέση των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα μπορούμε να υποστηρίξουμε. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερο τις δυνατότητες για ε, περισσότερη νομιμοποίηση των ε, εθνικών κοινοβουλίων. Οι εθνικές συνελεύσεις, για παράδειγμα, λέγεται ότι θα πρέπει να είναι ο χώρος όπου γίνεται η αυτοαξιολόγηση όσον αφορά το κράτος δικαίου. Αυτό είναι πολύ σημαντική πτυχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμα. Είμαι πεπισμένος ότι πολλά εξαρτώνται από το πώς οργανώνονται μόνα τους τα εθνικά κοινοβούλια, πώς αναπτύσσουν μηχανισμούς ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ευρωπαϊκή πολιτική. θα πρέπει να έχουμε μία θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με ελάχιστες μεταρρυθμίσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία χειρονομία και θα αποτελούσε κίνητρο για τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now... Σας ευχαριστώ. Σελίμοβιτς από την Άλντε, σκιώδης Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ράντζελ για την έκθεσή του. Συμφωνούμε όσον αφορά την ανάγκη απλούστευσης. Δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα είναι εύκολο. Διότι υπάρχουν εδώ δύο εξουσίες, τα Εθνικά Κοινοβούλια από τη μία που έχουν εκχωρήσει κάποιες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη έχουν εκλέξει και εμάς ώστε να θεσπίζουμε τους νόμους με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά συμφωνώ κύριε Ράγχελ ότι θα πρέπει η κοινοβουλευτική γραμμή να ε, απλουστευτεί. θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα εθνικά κοινοβούλια με τον ίδιο τρόπο που τα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά ή τοπικά. Δεύτερον, στηρίζουμε την ιδέα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας που θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Σημειώνουμε ε, αυτά που έχει πει ο κύριος Μακρόν. Πιστεύουμε όμως ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν κανείς έχει πρόβλημα σε Περιφερειακό Κοινοβούλιο, συζητιέται εκεί. Ε, αν έχει κανείς πρόβλημα σε Εθνικό Κοινοβούλιο, θα συζητιέται ε, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την Ευρώπη, στο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Επίσης, όσον αφορά ε, το θέμα των, ε, της πρωτοβουλίας των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Κόκκινη κάρτα, συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο και η πορτοκαλή κάρτα μας έχει δείξει ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που έπρεπε. Επίσης, όσον αφορά ε, την ε, τροποποίηση της προθεσμίας των 8 εβδομάδων. Αυτό μπορεί να γίνει διότι δεν ε, εγγράφεται στη συνθήκη. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, να μην ζητήσουμε καμία αλλαγή που να απαιτεί τροποποίηση της συνθήκης. Θα υποβάλουμε τροπολογίες. Κύριε Σιγητά, σας ευχαριστούμε για την καλή δουλειά σας. Ευχαριστώ κύριε Σελίμοβιτς. Παίρνω εγώ το λόγο πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ράντζελ. Θα μιλήσω Ιταλικά. Ε, Για να τα πω και πιο γρήγορα. Η ουσία αυτού που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά την άποψή μου αυτή η έκθεση γεννάται αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μια κρίση νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την άποψή μου θα πρέπει να προσθέσουμε και μια κρίση νομιμοποίησης των κρατών εθνών και επομένως το συζητήσαμε και στη συνεδρίαση των σκιωτών εισηγητών. Κατά την άποψή μου η ίδια η επικουρικότητα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί κατά κάποιο τρόπο, να διευκρινιστεί, να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει αυτή η διπλή κρίση και ε, να αναφέρουμε και τη σημασία που έχει η επικουρικότητα προς τα κάτω, όχι μόνο προς την κορυφή, αλλά και προς τις περιφερειακές εξουσίες ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά την ε, πολυφωνία. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κύριος Ρανζέλ για τα χαρακτηριστικά των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι να υπάρχει και η διαφορετικότητα, η διαφοροποίηση, κάτι το οποίο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών δεν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τις συμβάσεις που προτείνει ο Μακρόν, ε, εκείνο που θα έχει ενδιαφέρον είναι να προσπαθήσουμε να μάθουμε και λίγα περισσότερο, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει επακριβώς ε, ε, περί τίνος πρόκειται σε αυτή την πρόταση. Τελείωσα εγώ, θα είχα κι άλλα να πω, αλλά θα σεβαστώ το χρόνο και τώρα να δώσω το λόγο στον Μαξ Άντερσον. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που περιλαμβάνει πολλά καλά στοιχεία. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να σας πω πώς με ικανοποιεί η ιδέα μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας σύμβασης να έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τις 8 εβδομάδες και να δώσουμε κάτι το οποίο θα είναι πιο λογικό ως προθεσμία, χωρίς να χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό και μπορώ, μπορώ να συνταχθώ με την πρόταση αυτή. Επίσης, η ιδέα της χρήσης της πράσινης κάρτας είναι πολύ θετική. Αναρωτιέμαι όμως μήπως είναι αρκετά φιλόδοξη η πρόταση. Γιατί σε μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει βασικά προβλήματα, ακριβώς επειδή οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργούν το ίδιο καλά σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί δεν έχουν σχεδιαστεί με λαμβάνοντας υπόψη τις δημορφίες όλων των κρατών μελών. Οπότε, δεν θα έπρεπε εδώ τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να μπορούν να προτείνουν τροποποίησης κάποιες νομοθεσίας έτσι ώστε να ε, ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό γιατί τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συζητάνε το πώς θα επιλύονται τα διάφορα προβλήματα. Άρα θα έπρεπε λοιπόν να τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν μιλώ εδώ για δικαίωμα πρωτοβουλίας, τίποτα παρόμοιο, αλλά θα έπρεπε να τους επιτρέπετε να σχολιάσουν και να πούν αυτός ο κανόνας για μας δεν λειτουργεί. Σας παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν σα κάνει κόπο, φτιάξτε το. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί τμήμα της πράσινης κάρτας και υπάρχουν και άλλα θέματα στο οποίο θα μπορούσα να πω και νομίζω ότι σε μια επόμενη συνεδρίαση θα τα καταφέρω. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είμαι αντιπρόεδρος και έχω την αρμοδιότητα να παρακολουθώ τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η λέξη σχέσεις είναι εδώ όρος κλειδί. Εγώ δέχομαι τα τεχνικά ζητήματα όπως την επέκταση της προθεσμίας, την πράσινη κάρτα κτλ. Όμως σε κάποιο βαθμό αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εμβαθύνουμε στη σχέση αυτή σε πολιτικό επίπεδο, σε ε, κομματικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό το οποίο έχω ε, ανακαλύψει όσο έχω αυτό το ρόλο είναι ότι υπάρχει κάποιο είδος μία απολύτως υγιής ε, ανταγωνισμός και έλλειψης ε, εμπιστοσύνης μεταξύ ε, βουλευτών εθνικών και ευρωβουλευτών. Ε, και νομίζω ότι την ίδια δουλειά κάνουμε, απλώς καθόμαστε αλλού. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη συνθήκη για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Νομίζω ότι μετά το δημοψήφισμα στην ε, Αγγλία για να εγκαταλείψουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν έρθει πολλά κράτη-μέλη σε επαφή μαζί μας, επίσημα και ανεπίσημα για να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος μας ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις σχέσεις μας γιατί αν μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε πιστεύω πως θα έχουμε κάνει πολλά και θα ήθελα να συγχαρώ τον Πάολο Ραντζέλ για τις προσπάθειες που έκανε είναι σημαντική η δουλειά του και είναι και πολύ λεπτομερή η σύνταξη της έκθεσης Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Ραντζέλ Δύο λεπτά έχετε. Όχι, παραπάνω χρόνο χρειάζομαι. Ήδη μακρηγορήσατε πολύ κατά την παρουσίαση. Ε, ε, ε, Είμαι πολύ σύντομος, αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Στα όσα είπε η κυρία Περβάνς Περέες, ότι είναι περιγραφικά αυτά, όχι δεν είναι αλήθεια είναι απλώς προτάσεις. Σε όλη την έκθεση λέγεται ότι εάν τα εθνικά κοινοβούλια θέλουν πραγματικά να διαδραματίσουν ένα ρόλο και να μπορούν να ελέγξουν τις κυβερνήσεις και, τη σχέση, και να έχουν και σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αλλάξουν τον ιστορικό τους κανονισμό. Αλλά αυτό είναι κυρίαρχο δικαίωμα. Είναι το δικαίωμα της αυτοοργάνωσης, είναι το οργανιζασιόν σχεβάλτ του κάθε κοινοβουλίου. Και αυτό το χρησιμοποιώ απλώς για να πω ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της συμβολής των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι οι κανόνες θα πρέπει να προσαρμοστούν το Εθνικό Κοινοβούλιο για, τα Ευρωπαϊκό, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιστρόφως. Επίσης, δεν χρησιμοποιώ επακριβώς ε, την έκφραση πράσινη κάρτα για να πάω σε αυτό, προς αυτό που είπατε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι σωστές οι ενστάσεις σας, γι' αυτό ακριβώς και δεν ε, ακολουθώ τα όσα λέει ο κύριος Άντερσον, διότι υπάρχει... Ε, μια ισχυρή σκανδιναβική κοινοβουλευτική πίεση για το δικαίωμα ε, της ε, τροπολογίας αλλά το δικαίωμα της ε, τροπολογίας δεν είναι απλώς μετρήσιμο μπορείς να κάνεις το εξή. Μπορείς να δώσεις ε, εντολή στην κυβέρνησή σου, τη Σουαδική, τη Δανέζικη, τη Φιλανδική, για να ε, ε της δώσει εξουσία να τροποποιήσει κάποια πράγματα. Αλλά έχεις και δικαίωμα να ε, ζητήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει κάτι. Πρόκειται για ανεπίσημη εξουσία η οποία υπάρχει ήδη. Αλλά ε, εδώ πρέπει να είμαστε προσεπικτικοί. Δεν υπάρχει καμία αντιστροφή της κατάστασης, κανένα δικαίωμα τροποποίησης, κανένα δικαίωμα πρωτοβουλίας, αλλά με 4-5 κοινοβούλια μπορεί ίσως να ξεκινήσει μια διαδικασία ε, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει για να πει απλώς αν ε, συμφωνεί ή όχι και αν θα ακολουθήσει την πρόταση. Και εδώ και με αυτό θα ολοκληρώσω. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτω, γιατί αυτό γνωρίζω και από την πείρα μου με τη Μάρια Μαγκίνε, ότι εδώ είναι πολύ πιο σημαντική η δυναμική τη σχέση παρά οι τεχνικέ πτυχέ. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο στην ε, ε, αιτιολογική έκθεση υπάρχει ε, ένα όραμα του συγκεκριμένου ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιο το λέει αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό πιστεύω. Ε, παρεπιπτόντως όσον αφορά αυτό τον ανταγωνισμό, ο οποίος ε, θεωρώ ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα από ό,τι ε, στο παρελθόν. Χρησιμοποιώ μια έκφραση που χρησιμοποίησα στο παρελθόν. Είναι συνταγματική ε, Συνταγματικό φθόνο αυτό ο οποίο κυριαρχεί μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω όμω ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ όπω είπατε μετά τον Brexit. Ακόμα και πριν όμω είχαν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα και εδώ έχουμε μια σχέση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό οι πρωτοβουλίε, όπω η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, κάποιες ανεπίσημες πρωτοβουλίε, το ICM είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά σα ευχαριστώ την προσοχή, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολυφορία ε, και αναλογική εκπροσώπηση κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου. Και αυτό έχει σημασία, διότι ε, φέρνει την εσωτερική ποικιλομορφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό επιτρέπει και την διάσταση απόψεων και τη συγκερασμό απόψεων με τις ευρωπαϊκές οικογένειες και αυτό δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό πολιτικό πεδίο μάχης που είναι πολύ σημαντικό για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρανζέλ. Τέσσερα λεπτά μίλησα. Ευχαριστώ κύριε Ραντζέλ, σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Και τώρα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των τροπολογιών και της ψηφοφορίας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ε, στα αγγλικά αυτή τη συζήτηση. Το σχέδιο έκθεσης θα μεταφραστεί στις 19 Δεκεμβρίου. Άρα υπάρχουν δύο πιθανές εναλλακτικέ λύσεις. Η μία είναι να υπάρχει προθεσμία για τις τροπολογίες 12 ε, ε, ε, Δεκεμβρίου συγγνώμη, 20 Δεκεμβρίου ε, στις 5 η ώρα και μετά ψηφοφορία 20 με 22 Ιανουαρίου και το δεύτερο προθεσμία τροπολογιών 9 Ιανουαρίου του 2018 και ψηφοφορία 26-27 Φεβρουαρίου του 2018. Είναι σαφές ότι η πρώτη εναλλακτική λύση είναι πιο περιορισμένη Έχουμε δύο μέρες για τις τροπολογίες και ε, μετά η ψηφοφορία είναι λίγο πιο ομαλή. Εμένα μου φαίνεται λίγο καλύτερη, αλλά ε, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Εγώ προτιμώ τη δεύτερη, αλλά φυσικά αυτό απαιτεί και ε, θεσμική δράση. Αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, νομίζω ότι η Περβάνση είχε δίκιο ότι ήταν λίγο αισιόδοξη η προθεσμία του Ιανουαρίου. Το Φεβρουάριο είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα έχουμε το έγγραφο, μετά θα έχουμε τι μεταφράσει και θα υπάρχει και επαρκή χρόνο να υποβληθούν τροπολογίε. Αν είναι εφικτό ε, και το δεχτεί η διάσκεψη των Προέδρων, ε, τότε θα το περάσουμε εκεί. Εντάξει. Τότε οι ημερομηνίε είναι αυτέ. Εκτός μικροφώνου, κυρία Περές. 26-27 η ψηφοφορία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και γεια σας.